Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Άρχεται η συνεδρίασή μας. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Σεκέρσκι, κολλείεται για σήμερα και μου ζήτησε να προεδρεύσω εγώ σε αυτή την απογευματινή συνεδρίαση. Κάτι που θα κάνω με ιδιαίτερη χαρά. Θα ήθελα πρώτα να σας υπενθυμίσω όμως ότι η ψηφοφορία για τα μέτρα φυτοπροστασίας κατά των επιβλαβών οργανισμών που την είχαμε αναβάλει από την προηγούμενη μας συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο το πρωί η σχετική ψηφοφορία. Θα είναι το πρώτο σημείο της αυριανής ψηφοφορίας, το σημείο, νέο ναι, σημείο 4α. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να την εγκρίνουμε. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Επίσης να σας ενημερώσω ότι ε, γίνεται αναμετάδοση από το διαδίκτυο της συνεδρίασης μας απευθείας. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη ενημέρωση. Και επίσης αύριο εγώ, υποφαινόμενος και ο κύριος Μποβέ, σας προσκαλούμε για μια γευσηγνωσία των παράνομων ίνων. Κάπως παράδοξο και ιδιάζων που εκπρόσωπος της Επιτροπής Γεωργίας σας καλεί σε γευσηγνωσία παράνομων ίνων που θα γίνει αύριο από τις 12.30 το μεσημέρι στο μπαρ ε, Ζωζέ Φαντάλ, στο τρίτο όροφο του κτηρίου που βρισκόμαστε. Πρόκειται για ίνους ε, από ποικιλίε που είχαν αποσυρθεί από την αγορά στο παρελθόν. Αλλά βρήκαμε την ευκαιρία με τον κύριο Μπόβε να σας καλέσουμε σε αυτή τη γευσή γνωσία. Δεν μπορώ να σας εγγυθώ την ποιότητα, αλλά όσοι πιστοί προσέλθετε αύριο από τις 12.30 το μεσημέρι στην Πρεσερή, στον τρίτο όροφο του κτηρίου που βρισκόμαστε. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι έχουμε διερμηνεί από και προς 20 γλώσσες για τη συνεδρίασή μας αυτή. Και αυτά ως προς τα διαδικαστικά. περάσουμε τώρα στην δημόσια ακρόασή μας. Θα κρατήσει μέχρι τις 5 σήμερα το απόγευμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εφαρμογή της ενωσιακής Ομοθεσίας στον γεωργικό τομέα. Έχετε λάβει πληροφορίες για τη διοργάνωση της σχετικής δημόσιας ακρόσης που στόχο έχει μία σύγκριση και μία συζήτηση σε πολλά επίπεδα για την εφαρμογή της νοσιακής νομοθεσίας στον γεωργικό τομέα και μάλιστα σε όλα τα κράτη-μέλη. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε θέματα όπως η ευζοία, καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον. Θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στα διάφορα κράτη-μέλη που έχει η εφαρμογή της νομοθεσίας, το κόστος της και κρών στην γεωργία, η ποιότητα και η συσσόρευση κανόνων ό,τι αφορά την παραγωγικότητα των γεωργών και την ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά. Και στόχος μας στην ακρόαση είναι να προτείνουμε για κάποιες συστάσεις στους πολιτικούς ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στους εθνικούς πολιτικούς ηθήνοντες, προκειμένου να ε, θεσπιστούν ισότιμοι και δίκαιοι κανόνες για όλους τους ε, Ευρωπαίους γεωργούς. Καλέσαμε τέσσερις ε, εμπειρογνώμονες για να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Οι κανόνες είναι απλοί και διαφανείς. Θα δώσουμε από ένα δεκάλεπτο στον κάθε ομιλητή. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Ο πρώτος μας εμπειρογνώμονας είναι ο κύριος Νίλς Λίντμπερκ Μάτσεν. Είναι τιματάρχης στο Δανικό Συμβούλιο Γεωργίας και Τροφίμων. Θα μας μιλήσει για τις οικονομικές πτυχές της γεωργικής πολιτικής ή μάλλον περισσότερο για τι ισότιμε συνθήκε ανταγωνισμού και, και τη διαφάνεια, που είναι δύο αναπόσπαστα στοιχεία τη κοινή γεωργική πολιτική. Ο δεύτερο ε, εμπειρογνώμονά μα, που είναι ο κύριο Άνταλ Σαπατκάη, πρώην Γενικό Γραμματέα ε, τη Ένωση ε, Εργαζομένων στη Γεωργία από την Ουγγαρία, θα μα μιλήσει για τι οικονομικέ πτυχέ τη γεωργική πολιτική. Δηλαδή για το κόστο ισρών και παραγωγή εκρών στην φορολογική απλούστευση, απλοποίηση. Τρίτος ε, καλεσμένο είναι ο κύριο Άλμπερτ Γιάν Ματ, πρώην πρόεδρος Κοπακοζέκα και πρόεδρο τη LTO από τι κάτω που θα μα μιλήσει για τη σχέση μεταξύ τη γεωργική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γεωργικές πρακτικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο τέταρτο μα καλεσμένο είναι ο Ρόμπερτ Χόστ, ειδικευμένο οικονομολόγος στη χειροτροφία από το Ερευνητικό Ινστιτούτο γεωργικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Βάγγενιγκεν από τις κάτω χώρες και εκείνος θα μας μιλήσει για τους ότιμους ε, όρους ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή χειροτροφία. Δηλαδή θα συγκρίνει τις προδιαγραφές ε, σε θέματα ευζοίας και καλής μεταχείρισης και των περιβαλλοντικών κανόνων και προδιαγραφών. Για αυτά τα τέσσερα θέματα λοιπόν θα δώσω το λόγο διαδοχικά στους ε, εμπειρογνώμονές μας, στους καλεσμένους μας, πριν ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους συναδέλφους που θα σχολιάσουν. Πρώτος λοιπόν ο εισηγητής ε, Λίντσεν, Λίντμπεργκ Μάτσεν και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες όπως σας τους είχα παρουσιάσει. Κύριε Μάτσεν έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Είμαι από το Δανικό Συμβούλιο Γεωργίας και Τροφίμων που εκπροσωπεί τις εταιρείε τροφίμων και τους γεωργούς στη Δανία καθώς και τους κτηνοτρόφους. Συνδυάζουμε και τα δύο. Θα μιλήσω εν μέρη εκ μέρους τους και θέλω να προσφέρω και τη δική τους οπτική γωνία για την ε, Ευρώπη και το σύστημά της γενικότερα. Σε δύο βασικά σημεία θέλω να σταθώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την διερμηνία στα γαλλικά από ό,τι φαίνεται. Okay, thank you. Um, two main points Δύο κυρία σημεία. Πρώτα απ' όλα η σημασία των ισότομων κανόνων ανταγωνισμού με μια κοινή αγροτική πολιτική που σημαίνει και ενιαία αγορά. Και το άλλο είναι ο τρόπος τον οποίο θα καταλήξουμε εκεί, η διαφάνεια η οποία θα δώσει όχι μόνο στους γεωργούς και τους κοινοτρόφους, αλλά σε όλους τη δυνατότητα να συγκρίνουν τον τρόπο που γίνονται τα ίδια πράγματα σε άλλα κράτη-μέλη. Τι είναι ισότιμοι κανόνε ανταγωνισμού. Υπάρχουν πολλοί σχετικοί ορισμοί. Εγώ έχω δώσει εδώ ένα παράδειγμα. Αυτό που είναι πιο σκόπιμο για τη δική μας συζήτηση είναι από τη μια η εθνική νομοθεσία, θα μιλήσουμε αργότερα για φόρους. Είναι σημαντικό αυτό για να εξηγήσουμε τις διαφορές μεταξύ των κρατών. Υπάρχει τεράστια δυνατότητα ευελιξία στου ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή οδηγίε, και εκεί εντάσσεται και το θέμα για τη βασική γραμμή υπολογισμού όταν προβλέπεται νέα ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ποια είναι αυτή η βασική γραμμή βάσει της οποίας υπολογίζουμε την αμοιβή των γεωργών που ήδη έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Και τέλος, υπάρχει το θέμα της ε, πλημελούς υλοποίησης. Τα κράτη-μέλη που δεν καταφέρνουν να σεβαστούν πλήρως τους κανόνες. Ως προς την κοινή αγροτική πολιτική και το ισότιμους κανόνες λοιπόν. Η ενιαία αγορά είναι κέρια σημασίας αυτή θα εγγυηθεί την ύπαρξη την ίδια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Εάν δεν υπάρχει θα έχουμε μια κατακαιρματισμένη αγορά και θα ανταγωνιζόμαστε με ανισότιμους κανόνες. Ωστόσο, είναι δύσκολο και ήδη συζήτησα το τι γίνεται με τους πρωτοπόρους και τη συζήτηση περί της βασικής γραμμής του μέσου όρου. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν εγκρίνει κανόνε και διατάξει σε κάποιου τομεί και όταν γίνεται συζητήσει λόγω χάρη για τι κλιματικέ αλλαγέ, Είναι ένα καλό παράδειγμα. Επίση, πρέπει να δούμε το διοικητικό κόστο ε, κάθε φορά. Χρειάζεται περισσότερη απλούστευση για να μειωθεί το κόστο για του γεωργού Κάτι που θα ήταν τεράστια σημασία. Τέλος, η νομοθεσία πρέπει να προβλέπει αρκετή διαλλακτικότητα, αρκετή ευελιξία. Αυτό το είδαμε και στην τελευταία μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Και αυτό δεν είναι κάτι που εσεί ε, πρέπει να το δείτε εδώ κατά λεπτό σε αυτή τη διαφάνεια, δεν θέλω να δείξω όλε τι λεπτομέρειε και να τι εξηγήσω. Απλώ βλέπουμε πώ κατανέμονται οι άμεσε πληρωμέ σε επίπεδο κράτου μέλου. Οι διάφορε στήλε δείχνουν πώ αξιοποιούνται για το πρασίνισμα, για τη συνδεδεμένη βοήθεια, με το κόκκινο. Και βλέπουμε πόσε διαφορέ, τεράστιε διαφορέ υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Κάτι που το επιτρέπουν οι ίδιοι κανόνε, η ίδια νομοθεσία. Και μετά υπάρχει η άλλη όψη. Ορισμένα κάτι με, μελή πηγαίνουν πιο μακριά από ό,τι προβλέπουν οι οδηγίες ή οι κανονισμοί. Και βλέπουμε ότι κάποιοι καταβάλουν, καταβάλουν μεγαλύτερε προσπάθειε. Αυτό στη Δανία μα έχει απασχολήσει ιδιαίτερω. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε αυτέ τι αποκλήσει. Έχουμε ξεκινήσει κάποιε περίπτωση μελέτε και studies για να δούμε την υλοποίηση ορισμένων νομοθετημάτων, όπω για τα φωσβουργάλατα το περιβατάζω του χάλετα για τον, ε, ε, για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τη σχετική αποτίμηση, την οδηγία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την οδηγία για τα οικοσυστήματα, αυτά τα κοιτάξαμε για να δούμε αν μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος για τους δικούς μας τους γιώργους, τι πρόσθετο κόστος καταβάλουν ε, μεταξύ 400 και 600 εκατομμυρίων ήταν το αποτέλεσμα και οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλαπλοί. Είναι πιο αυστηρή η υλοποίηση της οδηγίας για τα αζωτούχα, για τα νητρικά άλατα και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσαμε για να πιέσουμε τη δανεική κυβέρνηση να αλλάξει τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί αυτό το νομοθέτημα ήταν αυτά τα στοιχεία που σας αναφέρω, δηλαδή τα στοιχεία με τα αριθμητικά ποσά ήταν πραγματικά ένας καλός μοχλός για να πιέσουμε την ε, ε, κυβέρνηση να κάνει κάτι γι' αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συζήτηση για την πολλαπλή συμμόρφωση και το πώς αυτή έχει υλοποιηθεί ως τώρα. Ακούσαμε φήμες, πάντοτε κυκλοφορούν πολλές φήμες για τους Γιώργους και τι κάνουν στην πράξη σε άλλα Πείσαμε λοιπόν το Δανικό Υπουργείο να κοιτάξει τι έχει γίνει σε γειτονικές χώρες και περιοχές. Κυρίως να δουν τους κανόνες, αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κάτι Το αποτέλεσμα ήταν ότι ήταν αδύνατο να δημορφώσουμε μια σαφή συνολική εικόνα. Το αποτέλεσμα ήταν η πόνοια μεταξύ των γεωργών ότι δεν του ενημερώνουμε πλήρω. Γιατί δεν μα ενημερώνετε πλήρω για αυτά που γίνονται στα αλλα κατημέλη. ήταν η απορία του. Και σκέφτονται ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, ότι κάποιο λάκκο έχει φάδα και ότι του το κρύβουμε. Υπήρχε λοιπόν μια υποψία για κάτι που δεν πήγαινε καλά εδώ. Αυτό που αποκομίσαμε ως δίδαγμα είναι Άλλα κάτι μέλη. Μοιάζει Ε, μοιάζει να τα πηγαίνουν καλύτερα στην πολλαπλή συμμόρφωση ε, και αυτό ήταν μια πληροφορία που μας ενδιαφέρει πολύ σε επίπεδο κυβερνητικό για να δημορφώσουμε την νομοθεσία μας. τι μας δείχνει αυτό, πού μας ε, φέρνει. Ότι έχοντας πληροφορίες και στοιχεία, αυξάνοντας το βαθμό διαφάνειας, θα έχουμε καλύτερα επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε ε, αυτό που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή θα έχουμε έναν καλύτερο τρόπο να μεταφέρουμε τις βέλτιστες πρακτικές από το ένα κράτος, από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Και όπως βλέπουμε θα αυξηθεί και η αξιοπιστία των ε, νομοθετημάτων, των κανονισμών και οδηγιών περί γεωργίας, με τις πληρωμές, με, το πρασίνισμα ή την ανάπτυξη της πέθρου ή την πολλαπλή συμμόρφωση. Αν γνωρίζουν οι γεωργοί τι συμβαίνει γύρω τους, θα έχουν και περισσότερη εμπιστοσύνη. Και είναι σημαντικό να δούμε και τις συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζονται. Όχι μόνο τι λέει ο νόμος, αλλά τι γίνεται στην πράξη στα ίδια τα αγροκτήματα και τι εκμεταλλεύσει. Η συγκεκριμένη μας πρόταση θα ήταν να έχουμε ένα βαθμολογικό πίνακα για την κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να μπορούν οι γεωργοί να συγκρίνουν ευκολότερα το τι συμβαίνει από το ένα κάτω στο άλλο και να διευκολύνουμε κατά την όλη συζήτηση για το πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερους, περισσότερο ισότιμους κανόνες. Για να ανακεφαλαιώσω, βασικό επιχείρημα για να έχουμε ισότιμους κανόνες είναι ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε μια κοινή αγροτική πολιτική που να λειτουργεί ως κοινή πραγματικά πολιτική. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους ισότιμους κανόνες για να έχουμε δικαιότερο ανταγωνισμό μεταξύ των γεωργών των διαφόρων χωρών. Εάν η διαφάνεια ε, δοθεί στους γεωργούς αν του αντιμετωπίσουμε δηλαδή με διαφάνεια, θα έχουν και οι ίδιοι μεγαλύτερη πίστη στην κοινή αγροτική πολιτική, γιατί θα διαθέτουν τι πληροφορίε που μπορούν οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν μέσω των ε, Υπουργείων ή στι συζητήσει τους με την Επιτροπή ή στις συζητήσει με εσά, μέλη αυτή τη Επιτροπής. Οπότε, θα ήταν ένα, ένας τρόπος να υποστηρίξουμε την καλύτερη νομοθεσία, να την προκαλέσουμε, αλλά κυρίως να διαλύσουμε και κάποιους μύθους που κυκλοφορούν. Δηλαδή, να μην νομίζουμε ότι όλα τα κάνουμε εμεί καλύτερα, αλλά έχοντα όλε τις απαραίτητε πληροφορίες να έχουμε μια πιο ε, τεκμηριωμένη συζήτηση για το όλο θέμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα τον άλλο ομιλητή. Κύριο Σάνταλ Σαμπαλκάη από την Ουγγαρία. Περιμένουμε να καθίσει θέση του. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θα συνεχίσω στα ουγγρικά την παρουσίασή μου. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ρίξουμε μια ματιά στην ε, παραγωγή, στα προϊόντα και στην ε, φορολογική αντιμετώπιση. Ο τίτλος της παρουσίασής μου είναι η θέσεις με την εξέλιξη των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία. Εγώ θα επικεντρωθώ στα οικονομικού περισσότερο χαρακτήρα ζητήματα στην παρουσίασή μου. Είδαμε αρκετέ ε, τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλαγές που αντιμετωπίζει ο παραγωγός και οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο, στον προσδορισμό των τιμών και τη σύνθεσή τους δύο χρόνια τώρα γίνεται μείωση της τιμής των, των τιμών των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας με σταθεροποίηση σε επίπεδα χαμηλότερα από ό,τι πριν, πριν από 2,5 χρόνια το ένα λίτρο κόστιζε 1,5 ευρώ. Στην Ουγγαρία τώρα κοστίζει ένα ευρώ λίτρο καυσίμου, έτσι έχει καμφθεί και η και ο πληθωρισμός από το 0,5 έχουμε ένα 0,1 περίπου. Και αυτό βέβαια βοηθάει την ε, προμήθεια σε προϊόντα ενεργειακά, πράγμα το οποίο βοηθάει ιδιαίτερα το μεγάλο ποσοστό ε, πολιτών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, που 25 με 30% είναι σε συνθήκες πολύ δύσκολες ε, και για το 2015 είχαμε 7,5 ευρώ κόστος ε, εργατικού δυναμικού, πολύ χαμηλό δηλαδή, πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 25 ευρώ και αντίστοιχα έχω ένα, μέσο όρο ε, εισοδήματος το μήνα, ελάχιστο μισθού δηλαδή, στο Βέλγιο 300, 1502 ευρώ, στην Ουγγαρία 333 ευρώ, ενώ στην Τσεχία 332 ευρώ. Έχουμε λοιπόν διάφορα χαρακτηριστικά, ευνοϊκά χαρακτηριστικά της γεωργίας. Από το 2010 προσπαθούμε να αποκομίσουμε με τα μέτρα της κυβέρνησης των δυνατόν περισσότερα ωφέλη. Έχουν ε, ενισχυθεί λοιπόν οι εργασίες στην Ήπεθρο, έχουν ενισχυθεί θέσεις εργασίας στην Ήπεθρο και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αποτέλεσμα τα κόμμα δεν είναι ορατά μένα, αλλά υπάρχει ε, ως, ένα, ως φαινόμενο ξεκάθαρο εδώ και καιρό η συγκέντρωση των νέων κυρίων στα αστικά κέντρα και η έξοδος δηλαδή από την ε, Ήπεθρο, η φυγή από την Ήπεθρο με την αστιφιλία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η συγκέντρωση σε μεγάλες ζωικές εκμεταλλεύσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση που έχει δημόσια γη να πουλήσει, την πουλάει, την πουλάει όμως στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί ε, και το εμπάρκο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρουσίας που ε, βρίσκονται ως υπόβαθρο στα προβλήματα όλα αυτά. Η, η κατανάλωση τρόφιμα έχει μειωθεί και λόγω των δημογραφικών τάσεων, των μειωμένων δημογραφικών τάσεων. Και όλα αυτά παρουσιάζουν σαν γενική εικόνα μια ευνή διαπτώση των τιμών των ε, τροφίμων, των γεωργών προϊόντων ως τροφίμων, ε, λόγω και της μείωσης εσωτερικής κατανάλωσης και της εξωτερικής ζήτησης. Έχουμε λοιπόν τις εξής, ε, τους εξής κινδύνους, με χαμηλότερη τιμή που καταβάλλεται στον παραγωγό, τιμή που μπορεί να είναι χαμηλότερη από το κόστος, λόγω της ε, πλεονάουσας προσφοράς και από την άλλη για τον καταναλωτή αυτό σημαίνει και στασιμότητα τιμών σε προηγου... ότι στασιμότητα τιμών σε επίπεδα προηγούμενων ετών ε, πιο ε, οικονομική βέβαια τιμή για τον καταναλωτή φαινόμενο το οποίο δεν χαρακτηρίζει μόνο την Ουγγαρία αλλά φαντάζομαι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν δούμε δύο ιδιαίτερους τομείς που έχουν προβλήματα, όπως όλοι βέβαια, δυσκολίες στην προσαρμογή, στην παραγωγή του χειρίου κρέατος, γιατί θα πάρω έναν, ως έναν αυτόν τον τομέα. Έχουμε χαμηλότερη παραγωγή. Οι παράγοντες αγοράς ε, διαμαρτύρονται για την ε, ε, για τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχει να κάνει και με φοροαποφυγή, αποφυγή καταβολής ΦΠΑ τουλάχιστον από μια μαύρη ή γκρίζα αγορά ε, και έτσι αυτό είναι εις βάρος του ε, ευσυνείδητου και έντιμου παραγωγού. Αυτό έχει να κάνει και με τα... με τη φορολογία αυτή σχετική με τα σφάγια που έχει αλλάξει. Επίσης, σε σχέση με το γάλα, ξέρουμε ότι το γάλα είναι ένα προϊόν ευπαθές, ιδιαίτερα κατά τη μεταφορά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν αρκετοί μηχανισμοί διαχείρισης των πλεονασμάτων, ρύθμισης της αγοράς. Τώρα έχουμε λοιπόν μείωση της, ε, του κόστους ε, της ε, διακίνησης του εξωτερικό της εξαγωγής επομένως ε, χαμηλότερες τιμές και ίσως αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Προτείνουν η παραγωγή γάλακτος ε, να μειωθεί ο φόρος για το ρευστό γάλα από το 25% στο 5% ΦΠΑ. Αυτό όμως δεν έχει γίνει δικτό. Υπάρχει σέμενο κρέας λιγότερο, φθηνότερο γάλα συγγνώμη, ε, γιατί δεν πληρώνει φόρο. Οι ειδικοί επίσης ε, λένε ότι υπάρχει και ένα είδος εκτελεστών του γάλακτος, ε, εντολοδόχων κυβερνήσεων που επιβάλλουν την επιβολή κάποιων φόρων. Νομίζω ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να είχαμε ε, και μείωση του ΦΠΑ στο γάλα όπως και στο χείριο κρέας. Για τα ζητήματα λοιπόν αυτά χείριο κρέατος και το γαλακτοκομικών παραγωμένου γάλακτος, ε, συνέπεια ε, απόρρια της επιβολής όρων περί ευημερίας των ζώων νομίζω ότι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σε μεγάλο βαθμό την, μείωση, την αύξηση του κόστους και ίσως θα έπρεπε να εξασφαλιστούν όροι πιο ευέλικτοι για τον ε, παραγωγό που εφαρμόζει την νομοθεσία αυτή από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, κινούμεθα... Έχουμε λοιπόν ένα φαινόμενο υπερπληθώρας από το 2009 στην Ουγγαρία. Η διαφορά μεταξύ κόστους και τιμης πολισεως πωλήσεως μειώνεται μεταξύ 2010-2015 η Γενική Γραμματεία Γεωργίας δημοσίευσε το 2015 ένα, μία μελέτη ανάλυσης ε, του τομέα γάλακτος και του χειρίου κρέατος για τη Γαλλία με προτάσεις εναλλακτική διαχείρισης της κρίσεως ε, δυνάμει κάποιων πιθανών σενάριων, υποθέσεων. Νομίζω ότι οι στατιστικές που έχουμε μπορούν να δώσουν ενδείξεις για κρίσεις. Έχουμε συγκριτικά στοιχεία που μας δείχνουν ότι το Νοέμβριο 2013 και μέχρι το Μάρτιο του 2016 η εξέλιξη είναι η εξή. Γαλλία με 24,4%, Ουγγαρία 30%, ε, Σλοβακία 24,2%, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 28,9%. Όλα αυτά σε αρνητικές τάσεις. Στις τιμές του γάλακτος. Φαίνεται ότι η παραγωγή γάλακτος θα αυξηθεί κατά 1% από ό,τι λένε οι και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί η παραγωγή. Ως ενδιάμεσο όμως μέτρο θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα αποθέματα γάλακτος σε σκόνη και βουτύρου. Έχουν αναλυφθεί κάποια μέτρα για τον περιορισμό κατά 3% της ε, παραγωγής γάλακτος μέχρι το καλοκαίρι. Και μια και δεν έχω χρόνο θα συντομεύω. και θα αφήσω ένα μεγάλο κομμάτι της παρουσίασής μου για να φτάσω στο τέλος, στο κομμάτι που αφορά τις γεωργικές αγορές και τις προοπτικές τους και τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις, γιατί πάντα έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση ε, αμφίροπη, το βλέπουμε και από τη γαλλική μελέτη. Είναι σαφές νομίζω, όταν εξετάζουμε τα στατιστικά δεδομένα και τις τάσεις, είναι πιθανότατο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρειαστεί να αναλάβει μέτρα παρέμβαση. Αυτά και για τον αλλακτοκομικό και για τον τομέα του χείριου κρέατος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στον τρίτο μας εμπειρογνώμονα, τον τρίτο καλεσμένο, Αφήνουμε λίγο χρόνο στον καλεσμένο μας να λάβει θέση. Δεν ακούγεται από το μικρόφωνο δυστυχώς. Χαίρομαι που ξανάρχομαι. Βλέπω παλιά, παλιούς γνώριμους, τον κύριο Ντές, τον κύριο Δεγκάστρο και νέα μέλη, την κυρία Σρέιερ, τον κύριο Γιάνν Χάιτεμα. Νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Θα συνεχίσω την ομιλία μου στα Ολλανδικά. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την οργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης για τους ισότιμους όρους αγωνισμού, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος για τους γεωργούς ε, και τους καλλιεργητές. Το θέμα δεν είναι τόσο οι τιμές όσο οι κανόνες του παιχνιδιού. Και αν δεν σεβαστούμε αυτούς τους κανόνες, η κρίση δυστυχώς θα επιδεινωθεί. Αυτό ισχύει για τη γεωργία, την αναπορκυπευτική, τη χειροτροφία Ε, και υπάρχει διαφορετικό επίπεδο συμμόρφωσης ε, μεταξύ των κρατών μελών. Πέρυσι είχαμε μια πολύ ε, σφοδρή συζήτηση στην κόπα Κοζέκα και βρέθηκαν τελικά 500 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε τους γεωργούς και κυπουρούς στην Ευρώπη να ανταπεξέλθουν στην κρίση. Έχουν περάσει 9 μήνες και 60% των κονδυλίων αυτών δεν έχουν εκδομηθεί ακόμη και μένουν πολλά φρούτα και λαχανικά αναξιοποιητά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους και να αξιοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, διαπιστώνουμε ότι για πολλούς τομείς έχουμε τις ίδιες οδηγίες, αλλά τις εφαρμόζουμε με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, για τα φυτοφάρμακα, για τα εντομοκτώνα. Ο βαθμός συμμόρφωσης εξετάται από τη χώρα. Ε, σε μία συνάντηση πρόσφατη στην ΚΟΠΑ, ένας Γάλλος συνάδελφος επισήμανε την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των Γεωργών και των Κυπουρών για να ανταπεξέλθουν από κοινό στην κρίση. Στις κάτω χώρες πληρώνεται για δίζελ 1,20 το λίτρο. Αλλά στις γειτονικέ χώρες οι τιμές είναι χαμηλότερες και μεγάλες διαφορές υπάρχουν από τη μία χώρα στην άλλη. Επίσης, το θέμα της πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα, τις εξαγωγές. Οι γεωργοί αναλαμβάνουν το πλήρες κόστος της πιστοποίησης, μέχρι και 15.000 ευρώ ανά, ανά χειροτρόφο για παράδειγμα. Αλλά βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστιες διαφορές μεταξύ γεωργών και κυπουρών στα διάφορα κράτη-μέλη. Και μπορεί η φορολογία να μην είναι κοινοτική αρμοδιότητα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού και εξασφάλισης ισότιμων συνθηκών και κανόνων. Οπότε θα πρέπει να το συζητήσει αυτό το Συμβούλιο Γεωργίας. Την περασμένη φορά το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση της κρίσης και το ποσό που θα πρέπει να αφιερωθεί σε αυτό. Και είπαμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί το κονδύλιο σε 15.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση. Αλλά τα κράτη-μέλη θα κρίνουν πώς θα εφαρμόσουν το μέτρο. Αλλά τα κονδύλια που χρειάζονται είναι πολλά. Και δεν θα είναι αποτελεσματικά αν δεν έχουμε ισότιμού όρου ανταγωνισμού. Μόνο εσεί μπορείτε να απευθύνετε έκκληση στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λιάνουν αυτέ τι διαφορέ και τι αδικίες. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η άνηση κατάσταση στο μέλλον και οι διακρίσει, δεν πρόκειται να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, η ισοτιμία. Είναι απαράδεκτες αυτές οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε τόσο σημαντικά θέματα. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου. Θα πρέπει να μειωθούν. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση ενίσχυσης της τοπικής γεωργίας και αυτό είναι σημαντικό, ειδικά για θέματα ποιότητα. Αλλά υπάρχει και το θέμα τη σήμανση σε εθνικό επίπεδο. Γιατί στα σύνορα μιλούμε για κάποια κοινά πρότυπα και προδιαγραφές και ίσως υπάρχει μια ελάχιστη τιμή που εφαρμόζεται, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε τα στρεβλωτικά αποτελέσματα μεταξύ των διαφόρων τελεστών στον κλάδο, στο Γεωργία και την απορροκυβευτική. Και μάλιστα στις κάτω χώρες οι γεωργικές ζώνες είναι πολύ κοντά στα σύνορα και υπάρχουν κινήσεις διασυνοριακές. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι από την άλλη πλευρά των σύνορων και να εμπίπτει στην τοπική οικονομία και στην βραχία λυσίδα ανεφοδιασμού. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο των αποφάσεων στους γεωργούς και τους καλλιεργητές οπωροκυπευτικών και στις όμορες ζώνες. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να θέσετε το ζήτημα και σε επίπεδο Συμβουλίου, γιατί 60% των 500 εκατομμυρίων που ε, προβλέπονται για την αντιμετώπιση κρίσης δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμη και δεν έχουν αξιοποιηθεί. Επίσης, ε, σίγουρα θα υπάρχει περιθώριο λιγμών σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των ισότιμων όρων και κανόνων του ανταγωνισμού. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στο κόστος των ισρώων. Και από τη στιγμή που μιλάμε για κοινή γεωρική πολιτική θα πρέπει να έχουμε ίδιους κανόνες. Και μάλιστα η Γεωργία και η Κυπουρή παράγουν το σημαντικότερο προϊόν για μας, το τα σημαντικότερα αγαθά. Γι' αυτό αξίζουν οι μεταχείρισης. Να, να μην αντιμετωπίζουμε με δίκαιο τρόπο τους ποδοσφαιριστές μας που μπορούν να παίζουν οπουδήποτε σε οποιαδήποτε ομάδα θέλουν στην Ευρώπη και να εφαρμόζουμε διακρίσεις για τους γεωργούς μας που παράγουν ένα τόσο πολύτιμο αγαθό. Από λοιπόν που δεν επιτρέπονται διακρίσει στον αθλητισμό, είναι απαράδεκτο να εξακολουθούν να υπάρχουν στη γεωργία και την, τον οποροκυπευτικό κλάδο. Ευχαριστώ. Merci. <coughs> Merci à vous, Ευχαριστώ πολύ. Euh, ευχαριστώ και περνάμε στον τέταρτο εμπειρογνώμονά μας. Θα είχατε την καλοσύνη κύριε Χώστα να μας ε, παρουσιάσετε την, ο... την ομιλία σας. Quelques secondes de, de patience le temps que le PowerPoint s'ouvre. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σα και θα σα μιλήσω για του ισότιμου κανόνε ανταγωνισμού στη χειροτροφία. Ιδιαίτερο. Και θα κάνουμε συγκρίσει ε, σε προδιαγραφέ ευζοία ε, και περιβαλλοντικέ και, το... και τι συνέπειε στο κόστο. Ξεκινούμε από την πυραμίδα. Βλέπετε τη βάση που είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για όλες τις χώρες μέλη. Αλλά τις ίδιες οδηγίες τα κράτη-μέλη τις ερμηνεύουν διαφορετικά. Πιο πάνω στην πυραμίδα έχουμε τις εθνικές προσθήκες, έχουμε τους εθνικούς συμπληρωματικούς κανόνες, τους εσωτερικούς και τέλος την κορυφή της πυραμίδας που είναι η εφαρμογή. Γι' αυτό δεν θα μιλήσω. Να σας αναφέρω μερικέ οδηγίες. Έχουμε την οδηγία για τα νητρικά άλατα πρώτον, μετά τα ανώτατα, ε, σε εθνικές εκπομπές ε, και άλλες που δεν σας αναφέρω, για τη μεταφορά, τη σφαγή των ζώων, τις σχετικές οδηγίες. Έχουμε όμως και συστάσεις και φιλοδοξίες για τη χρήση των αντιβιωτικών, ε, για, τις, ε, για τους ευνοχισμούς και τώρα έρχομαι στις ε, εθνικές ερμηνείες που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Θα σας αναφέρω μερικές από αυτές τις ερμηνείες. Σε ό,τι αφορά τις ε, περιβαλλοντικές άδειες, έχουμε διαφορετικές απαιτήσει και προδιαγραφές μεταξύ των κρατών μελών και έχουμε και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, προθεσμίες για την υποβολή αίτησης και τη λήψη της άδεια. Διαφορές έχουμε ακόμη και σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, ε, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν με διαφορετικές απαιτήσεις για το πότε χρειάζεται μια τέτοια μελέτη πτώσεων. Σε ό,τι αφορά την υποβολή ε, αιτήσεων για τη χρήση νητρικών και φωσφορούχων αλάτων, επίσης υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν εποχιακές διαφορές, ε, υπάρχουν διαφορές για την επεξεργασία της κοπριάς μεταξύ των κρατών μελών, εφαρμογή των εξαιρέσεων και εκεί υπάρχουν διαφορές. Και όλα αυτά αφορούν την ε, εθνική ερμηνεία της ενωσιακής νομοθεσίας, που εν μέρη αφορά και ε, έσχεται, έχει σχέση και με την πυκνότητα των, ε, του πληθυσμού. Για παράδειγμα, στη Δανία έχουμε πρόταση για μείωση των αριθμών ε, των κοπαδιών των χείρων. Σε ό,τι αφορά την αμμονία, μιλούμε για τις καλύτερες ε, ε επιτρε... ε, διαθέσιμες τεχνικές. Επίσης, τα επίπεδα μείωσης που θα πρέπει να επιτύχουμε στις εκπομπές αμμονίας. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιτυχάνονται αυτές οι μειώσεις ε, είναι διαφορετικέ. Επίση, ό,τι αφορά την επιθεώρηση των ε, ζωντανών ζώων, αναφέρθηκαν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι είναι πολύ διαφορετικοί από χώρα σε χώρα. Σε κάτω χώρε, ένα κτηνίατρο θα πρέπει να είναι ε, παρόν στην χειροτροφική μονάδα. Σε άλλε χώρε δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το κόστο είναι διαφορετικό. Σε ορισμένε χώρε το κόστο το αναλαμβάνει η χώρα και σε άλλε όχι. Επίση, ε, έχουμε τη μεταφορά ε, του κόστους ε, είναι 15 σέντα ένα χειρίδιο και ένα ε, ευρώ και κάτι όταν πρόκειται για εξαγωγή. Ακόμη, εξαγωγή, αν και η εξαγωγή αφορά μεταφορά σε 100-200 χιλιόμετρα εκτός της χώρας για να σφαγεί σε άλλο σφαγείο. Οπότε υπάρχουν μεγάλες διαφορές στους κτηνιατρικούς ελέγχους για την εξαγωγή των σφαγείων. Επίσης έχουμε τις εθνικές συμπληρωματικές διατάξεις. Έχουμε ένα ενδεικτικό κατάλογο εδώ. Καταρχήν, ε, το χώρο διαβίωσης 0,65 ε, ε, τετραγωνικά μέτρα λέει οδηγία για χειρίδια πάχυνσης μέχρι 110 κιλά σε ό,τι αφορά τον ελεύθερο χώρο διαβίωσης. 0,75 τετραγωνικά μέτρα είναι στην Γερμανία, 0,8 στις κάτω χώρες και στην Ελβετία πολύ λιγότερο. Βλέπετε, ανάλογα τη διαφορά του ε, χώρου είναι σημαντικό και το κόστος. Επίσης, για τις ε, χειρομητέρες που, που κυοφορούν, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου πρέπει να είναι 2,25 και 1,64 ε, για, για τα θηλυκά χειρίδια, τα μικρότερα. Επίσης, λέμε ότι η διαβίωση θα πρέπει να γίνεται σε ομάδες και τέσσερις, ε, με, τέσσερις εβδομάδες μετά την αλοχία στις ε, κάτω χώρες είναι τέσσερις μετά την τεχνική ε, σπερματέχηση. Σε άλλες χώρες είναι διαφορετική προθεσμία. Επίσης, ό,τι αφορά τον ελεύθερο χώρο δαπέδου, ε, τα χειρίδια πάχησης στις κάτω χώρες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 40% ελεύθερο χώρο δαπέδου, κάτι που δεν απαιτείται στην οδηγία. Και επίσης υπάρχουν διαφορές στον ορισμό. Τι εστί ελεύθερος χώρος δαπέδου, ε, 5 με 15% ελεύθερος χώρος και εκεί υπάρχει διαφορά μεταξύ των μελών. Σε ό,τι αφορά τους ακροτηριασμού η οδηγία προβλέπει ε, για τα χειρίδια διαφορετικού τρόπου έχουμε απαγορεύσει στη Σουηδία, Φιλανδία, Λιθουανία για ορισμενε περιπτωσει επιση η πικρότητα στη μεταφορά με φορτηγό. Τέσσερα χειρίδια είναι ο κανόνας μέχρι 100 κιλά, αλλά πάλι υπάρχουν διαφορέ. Στη Δανία υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνε για μεταφορά μεγάλων αποστάσεων. Στη Γερμανία υπάρχουν διαφορετικέ διατάξει για τι εγχώριε μεταφορέ. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του σανού. στη Σουηδία έχουμε υψηλό επίπεδο καλή μεταχείριση και αψοεία. Απαιτείται εξασφάλιση σανού για όλα τα, χειρινά, για όλα τα χειρίδια του κοπαδιού. Βλέπετε λοιπόν πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι εθνικές προσθήκες. Επίσης έχουμε μία επιλογή εθνικών μέτρων, τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Βλέπετε ότι στις κατοχώρες έχουμε 19 ε, λεπτά του κόστους, ε, συμμόρφωση με τους κανόνες, ε, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με την Ολλανδική ερμηνεία και τις εθνικές προσθήκες. Τα περισσότερα από τα 19 αυτά λεπτά του ευρώ αφορούν μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, ε, ε, χρήση της κοπριά και εκπομπές αμμονίας. 13 λεπτά συνολικά. Άλλες χώρες, ε, Γερμανία, Δανία, Πολωνία, Ισπανία, Γαλλία. Είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος βλέπετε. 7, 7, 8. Βέβαια, τι είναι 19 λεπτά. Αν πάτε σε ένα μαγαζί για να αγοράσετε ένα προϊόν, τίποτα. Αλλά 4 λεπτά είναι για έναν κτηνοτρόφο εισόδημα. Γιατί αν κάποιος ε, με από τη χειροτροφία και έχει ε, ακόμη και 4 λεπτά το θεωρεί εισόδημα, τα 19 λεπτά είναι πολύ μεγάλο ποσό. Επίσης έχουμε κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Έχουμε την κοινοτική νομοθεσία, αλλά επιπλέον έχουμε το λιανεμπόριο ή τους λιανεμπόρους, αλλά και άλλες αρχές που μπορούν να, δε, να θεσπίσουν τις δικές τους προδιαγραφές. Βλέπετε εδώ για Έχουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την Εθνική Νομοθεσία, την Ερμηνεία, τι συμπληρωματικέ εθνικέ διατάξει, αλλά έχουμε και του λιανεμπόρου που μπορούν να θεσπίσουν τι δικέ του ιδιωτικέ διατάξει και κάποιε ιδιωτικέ πρωτοβουλίε με σήματα, με, με μια ιδέα, με μια ορολογία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και αυτό είναι υπεράνω των ε, νομικών προδιαγραφών των νόμιμων συγγνώμη, προδιαγραφών. Οπότε όταν έχουμε κάποιες απαιτήσει που ξεπερνούν τις ε, ε, νόμιες προδιαγραφές, το κόστος το ε, φέρνουν κυρίως οι καταναλωτές. Και εδώ οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έχουν για τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις κάποιο ισότιμε συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά τις επιπλέον τέτοιες προδιαγραφές οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώσουν. Έχουμε λοιπόν το ένομο σύστημα και πέραν τούτου τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Και υπάρχει διάκριση μερικές φορές στις ε, απαιτήσει που έχουν οι συγκεκριμένοι λιανέμποροι. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε και με τις υπόλοιπες περιοχές ε, εκτός Ευρώπης. Ε, κάναμε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καν νομοθεσία για την ευζοία, για την καλή μεταχείριση των ζώων. Στηρίζονται σε βιομηχανικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές των λιανέμπορων και τις χρηστές γεωργικές πρακτικές. Και οι γεωργοί ε, στη χειροτροφία, για παράδειγμα, ασχολούνται με τις βιομηχανικές προδιαγραφές έχουν αντίστοιχε προδιαγραφέ ευζοία. Υπάρχουν κάποιε μικροδιαφορέ σε ό,τι αφορά την ομαδική διαβίωση για τι ε, κεοφορούσε χειρομητέρε, αλλά υπάρχει αυτό το σύστημα, ενώ στην Ευρώπη υιοθετούμε διαφορετική προσέγγιση με βάση την, εσωτερική, την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μετά έχουμε την εθνική ερμηνεία, τι συμπληρωματικέ εθνικέ διατάξει και επιπλέον έχουμε και τι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και προτείνω να περάσουμε στη συζήτηση αυτή αμέσω. Η Επιτροπή δεν θέλει να λάβει το λόγο το παρόν στάδιο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Λουαζού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται πως εγγυάται την ισότητα μεταξύ των κρατών μελών, αλλά εισάγει ένα σύστημα άδικο, άνισο, με έμφαση στην, στον ανταγωνισμό σε κάθε τομέα, με μια νέα σειρά κανόνων που σωρεύονται εδώ και δεκαετίες, δυσκολεύοντας όλο και περισσότερο τη δουλειά των γεωργών. Η προστασία του περιβάλλοντος βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η συσσόρευση ευρωπαϊκών κανόνων ε, σε, για τα κράτη-μέλη καθίσταται πλέον αφόρητη, ενώ γίνεται λόγος για απλούστευση τη ΠΑΚ εγώ που είμαι ο ίδιος γεωργό, όπως όλοι οι άλλοι γεωργοί, δεν βλέπω να έχει συμβεί τίποτε, θα έλεγα μάλλον ότι περιπλέκονται τα πράγματα. Το κόστος της εργασίας λοιπόν και όπως ξέρετε πολύ καλά η αμοιβόμενη εργασία που χρησιμοποιείται σε ορισμένε χώρε καθιστούν τελείω άνεσο τον ανταγωνισμό, καθώ και η άνεση εφαρμογή τη νομοθεσία τη σχετική με τα φυτογενή προϊόντα, ορισμένα εκ των οποίων είναι απαγορευμένα στη Γαλλία, όπως το τιμητοάτ, που θεωρείται καρκινογόνο, χρησιμοποιείται ως ε, φυτοπροστατευτικό στα κεράσια και καθώς δεν υπάρχει ε, νομοθεσία και μάλιστα θεωρείται ότι είναι και το μόνο που μπορεί να προστατεύσει το κεράσι, καθώς δεν υπάρχει πανευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, χρησιμοποιείται στις υπόλοιπες χώρες. Η ΕΦΣΑ, ε, σημειώνω, έχει δηλώσει ότι δεν έχει επαρκή στοιχεία για την γενίκευση της απαγόρευσης του συγκεκριμένου προϊόντος και άρα η Γαλλία είναι μόνη της στην απαγόρευση με συνέπεια φυσικά την αύξηση τη των κερασιών με δυσμενή για μας ανταγωνισμό. Αυτά ήταν ένα μικρό παράδειγμα της κατάστασης στην Ευρώπη. ευχαριστώ. Ο κύριος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη σημερινή εκδήλωση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την Επιτροπή μας να εξετάσουν όλες αυτές τις πτυχές. Για την νομοθεσία, επί ότι πρέπει να μεριμνήσουμε για όσο δυνατόν ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Πρέπει να κοιτάξουμε τις ε, διατάξεις και τον τρόπο που εφαρμόζονται αυτές στον οικονομικό, στο οικονομικό επίπεδο. Εγώ έχω πει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερη ε, διακύμανση με βάση το άρθρο 186, πρέπει τα 500 εκατομμύρια να διπλασιαστούν, διαρθρωτικά μέτρα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και χρειάζονται βέβαια υποστήριξη. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ώστε να ισότιμες ε, συνθήκες. Δεν θέλω λοιπόν να ρωτήσω ε, τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε κύριε Μάτ ως ε, μέτρα τα οποία μπορούν να έχουν έστω και είναι διαφορετικά ισο, ισοδύναμα συνέπειες στα κράτη-μέλη και αντίκτυπο. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα της ενίσχυσης των εισοδημάτων. Ο κύριος Δες, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τους τέσσερις ειδικού μας που ήρθαν να μας ενημερώσουν. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας ε, είπαν. Έχω κάποιες, ερωτήσει κάποιες ερωτήσεις και εγώ από πλευρά μου. Στην πρώτη τοποθέτηση έγινε λόγος για μεγάλη ευελιξία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η διατύπωση. Έχουμε να κάνουμε τεράστια στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα ως προς την υλοποίηση της γεωργικής μεταρρύθμισης και λόγω των υφισταμένων διαφορών μεταξύ των κρατών. Γι' αυτό λοιπόν... Θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε ίσως τόσο μεγάλες διαφορές ως προς τις πληρωμές των πρώτο πυλώνα μεταξύ κρατών μελών, αλλά έχουμε τεράστιες ε, διαφορές μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη και Κοιτάω προς τον πρόεδρο. Στη Γερμανία, Φερρυπίνα, έχουμε από 10 μέχρι 1000 ευρώ ε, πληρωμή ανά εκτάριο, ενίσχυση ανά εκτάριο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κοιτάξουμε και θέλω να σημειώσω. Μια και έγινε λόγο ότι τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα διαθέσιμα 500 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα ήταν καλύτερα αυτά τα 500 εκατομμύρια αντί να τα χρησιμοποιήσουμε ραντίζοντας με αυτά τα χρήματα δεξιά και αριστερά να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώση των αγορών γιατί έχουμε παραδείγματι ε, βούτυρο που έρχεται από την Ινδονησία στην Ευρώπη με πολύ χαμηλές τιμές και βεβαίως αν μπορούσαμε να σταθεροποιήσουμε τις αγορές θα μπορούσαμε να έχουμε ε, τεράστιο αντίκτυπο. Ιδιαίτερα δε με απασχολεί το γεγονός και αναφέρθηκε ότι λέμε στον Γεωργό πως μπορούν να ε, αφήνουν να εμποδίζουν κατά κάποιο τρόπο το, τα προϊόντα από τη μία χώρα στην άλλη και να μην φτάνουν αυτά έτσι στο ράφι του ε, σούπερ μάρκετ. Αν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν περιορισμοί ως προς την κυκλοφορία των γεωργικών προϊόντων από τη μία χώρα στην άλλη, τότε μπορούμε να ξεχάσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ε, από τη Γερμανία στην Ιταλία ή τη Γαλλία ή αντίστροφα δεν θα περνάνε τα προϊόντα και τότε δεν θα έχει κανένα νόημα να μιλούμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε είδαμε και ε, εχθές αυτά που συνέβησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι και πρέπει να τα φροντίσουμε αυτά, ιδιαίτερα δε στη γεωργική πολιτική. Oui, M. De Castro. Κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου τους εμπειρογνωμονές μας για τις τόσο ενδιαφέρουσες εισηγήσει τους και διαπιστώνω ότι υπάρχει έλλειψη ισοτιμίας κανόνων στα κράτη, μεταξύ των κρατομελών και αυτό μας οδηγεί σε έναν κίνδυνο που διαρκώς αυξάνεται επανεθνικοποίησης της αγροτικής πολιτικής. Όπως ήδη υπόθηκε από τους προλαλήσαντες, εμείς σημειώνουμε ότι υπάρχει κρίση το γαλακτοπαραγωγικό τομέα με πτώση τιμών 30% ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Νοέμβριο του 2013 ως σήμερα και δεν έχουμε αντιδράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχουμε βρει μια ευρωπαϊκή λύση σε όλα αυτά. Έχουμε εκχωρήσει την ευθύνη στα κράτη-μέλη και αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τέλει σε μεγάλο βαθμό αφοσιώθηκαν στην ανακατανομή μεταξύ των χωρών χωρίς καμία αποτελεσματικότητα. Και ακριβώς, όπως είπε και ο συνάδελφος Ντες, σε μεγάλο μέρος δεν έχουν δαπανηθεί και σωστά. Υπάρχει λοιπόν κινδύνος επανεθνικοποίησης των αγροτικών πολιτικών. Είναι πολύ υψηλό και δεν φαίνεται να βρίσκουμε λύση. Λύση στα προβλήματά μας. Μάλλον, καλό είναι να γυρίσουμε σε ευρωπαϊκέ πολιτικέ που να είναι λίγο αμεσότερε. Να μην εκχωρούν τόσε ευθύνε στα κρατη Η ευελιξία ε, κινδυνεύει να ε, φέρει μια ριζοσπαστική επανεθνικοποίηση των πολιτικών. Εδώ χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές αποκρίσεις και για να το πετύχουμε αυτό πραγματικά και σας παραπέμπω στην ε, ερώτηση του πρόεδρου Ματ. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση, να την κάνουμε ή απλώς είναι ένα σύνθημα διότι αν πραγματικά θέλουμε να την κάνουμε, πρέπει να βάλουμε κάτω και να εξετάσουμε τα νομοθετικά κείμενα. Αλλιώ παραμένει κάτι το τελείω φανταστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον εμπειρογνώμων από την Ουγγαρία σε ό,τι αφορά τα μέτρα μείωσης ε, του συντελεστή του ΦΠΑ. Τελικά τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν, απέφεραν καρπούς και η μείωση από 20% σε 5% αφορούν μόνο τα σφάγια, τα μισά σφάγια ή μειώθηκε ο ΦΠΑ και για το γάλα ή και για άλλες ε, γεωρικές παραγωγές ή μήπω ε, μόνο εξαιτία τη κρίση δύο αυτού του τομεί επιφέρατε μείωση του συντελεστού για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Σρέιερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ χρήσιμη και σκόπιμη αυτή η ακρόαση. Ήδη την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε για την κρίση στη Γεωργία. Τώρα πρέπει επιτέλους να λάβουμε δράση. Θα ήθελα να κάνω μια πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Ματ. Στις 7 Αυγούστου ξεκίνησε το εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Τώρα βλέπουμε τις επιπτώσεις. Ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με αυτά τα 500 εκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί δεν πρέπει να, να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα αυτά θα φτάσουν στα χέρια σου πραγματικά τα χρειάζονται. Διότι γιατί δεν δαπανώνται όπω θα έπρεπε. Αυτό εξαρτάται από ότι είναι απόφαση των κυβερνήσεων. Την περασμένη εβδομάδα, λόγω χάρη, οι χειροτρόφοι είπαν ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμα στου εκτροφεί βοηδών, λόγω χάρη. Και εάν δούμε τι γίνεται στη Γαλλία, την ε, Δανία ή το Βέλγιο, πραγματικά υπάρχουν διαφορές ε, στο πώς εφαρμόζονται οι κανόνες. Και μετά να δούμε και την πιστοποίηση. Οι πολίτες έχουν στείλει ε, χιλιάδες επί χιλιάδων mail γιατί θέλουν να μάθουν από πού φτάνουν τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν. Θέλουν να είναι σαφή η σήμανση πρώτα από μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να πολλούνται εύκολα ή να έχουν καλές πωλήσει. Είναι σημαντικό λοιπόν και οι γεωργοί να ξέρουν τι κανόνες πρέπει να τηρούν. Και τώρα μια ερώτηση προς τον δόκτορα Χώστε, ο οποίος μίλησε για το υψηλό κόστος των, ε, της παραγωγής χείριου κρέατος ε, στις κατοχώρες. Ε, ο Υπουργό Φαντάμ τη χώρα μα είπε ότι βεβαίω ε, έχουν γίνει υψηλέ επενδύσει για την ευζοία των ζώων και το περιβάλλον και την προστασία του δηλαδή, αλλά χρειαζόμαστε και κέρδο από όλα αυτά. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει και απόσβεση όλων αυτών των επενδύσεων. Αυτό δεν συμβαίνει όμω πάντοτε. Ξέχασα μια σημαντική ερώτηση. Σα παρακαλώ, Πρόεδρε, μπορώ. Ωραία. Ε, το Natura 2000 και η σχετική οδηγία για τα οικοσυστήματα. Εδώ έχουμε μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα ε, που καταρτίζει πολλές διαφορετικές περιοχές. Εδώ χρειάζονται κάποιοι συγκεκριμένοι προσανατολισμοί. Ήθελα λοιπόν να μου πει ο κύριος Ματ, θα ξέρετε ότι στις κάτω χώρες υπάρχουν απαλωτριώσεις, όχι μόνο στη δική μου την περιοχή, αλλά σε όλη τη χώρα. Ε, πρέπει και στις κάτω χώρες να φροντίσουμε οι προσανατολισμοί να ε, ακολουθούνται, αλλά όχι εις βάρος των ε, Ολλανδών ε, γεωργών, διότι αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε καν εκτροφής ε, βοηδών, ούτε παραγωγή γάλακτο στις κάτω χώρες. Κύριος Χάουσλινγκ. <clears throat> Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Με ξάφνιασε το γεγονό ότι το Front National είναι αυτό το οποίο διαμαρτύρεται που δεν έχουμε μια ενιαία πολιτική. Πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό το βρίσκω στη συζήτηση να ακούγεται ενώ γίνεται λόγος για πανεθνικοποιήσεις, για Brexit και για δεν ξέρω τι άλλες πολιτικές, ε, να βγαίνει το Front National και να αντιτίθεται στη μοναδική πολιτική, εθνική πολιτική που έχει η Γαλλία. Με βάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει σε πολλούς τομείς ακόμη να προχωρήσουμε προς την ενοποίηση, προς κοινά μέτρα. Έχουμε πάνω απ' όλα πρόβλημα στη ρηλοποίηση των υφισταμένων μέτρων. Υπάρχουν προβλήματα ως προδιαγραφές στις συνθήκες ε, εκτροφής των ζώων σε κλουβί ε, ή σε στρομνή για τους χείρους ε, βλέπουμε ότι δεν υλοποιείται με σωστό τρόπο η νομοθεσία. Άρα χρειάζεται να έχουμε βεβαίως με κάποιες διαφορές ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ε, κλιματολογικές ε, και τις κοινωνικές και τις εδαφικές ε, θα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει όμορφη εφαρμογή. Μπορεί στην Γερμανία ή την Ολλανδία να είναι μεγαλύτερες οι από ό,τι φερειπίν στην Ιρλανδία. Έχουμε εδώ άλλες προδιαγραφές ή μάλλον πρέπει να έχουμε διαφορετικές προδιαγραφές ε, φερειπίν σχετικές με την χρήση λιπασμάτων και το καθεξής ε, λόγω της πυκνότητας, διαφορετικής πυκνότητας του πληθυσμού των ζώων. Και πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να μας απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα της σήμανσης, της επισήμανσης των προϊόντων ανάλογα με το είδος της κτηνοτροφίας, της προέλευσής τους, ε, και χωρίς να έχουμε ενιαίες τιμές θέλουμε να έχουμε μια ενιαία επισήμανση ακριβώς για να μπορεί ο καταναλωτής και με βάση βέβαια την τιμή που θα του προσφέρεται να κάνει την επιλογή με το ε, λόγο γνώσεως. Νομίζω ότι μετά τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής δεν μπορεί κανεί να ισχυριστεί ότι έχουμε μεγαλύτερες ανισότητες. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον ε, να προσαρμόσουμε την επιδότηση επιφανείας, αναεπιφάνεια. Υπάρχει ασφαλώ ένα μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξία στο δεύτερο πυλώνα, αλλά προσπαθήσαμε νομίζω την προσαρμογή να την κάνουμε σε σχέση με τι επιδοτήσει, Δεν ξέρω αν οι δικοί μα θέλουν να απαντήσουν. Ευχαριστώ, Φερά. Ευχαριστώ. Ε, πραγματικά εξεπλάγει μια ναι, και για πρώτη φορά έχουμε μια πολιτική συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Ευνηδιάστηκα γιατί η Γεωργία δεν είναι ούτε της αριστεράς ούτε της δεξιάς. Και το να κρίνουν όπως ε, ο κύριος Δεκάστρο και ο κύριος Δες στην Ευρωπαϊκή κατάσταση, στην Ευρωπαϊ... την πολιτική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη μεταφέρουν στη Γεωργία νομίζω ότι είναι πολύ βαβιασμένο. Κύριε Ντάς, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την εσωτερική κατάσταση της αυστριακής πολιτικής. Και κύριε Ντεκάστρο, αν θέλετε ε, τα κράτη να μην επιλαμβάνονται πια των ε, γεωργικών θεμάτων, αλλά μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις τη για τη Γεωργία. Αν κάτι τέτοιο επιθυμείτε, δικαίωμά σας είναι να θέλετε να πολιτικοποιείτε την Επιτροπή Γεωργίας. Αλλά για πρώτη φορά έχουμε μια πολιτικάντικη ε, συζήτηση, μια πολιτικοποιημένη συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Ε, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι, ε, δεν αρμόζει και σίγουρα δεν μας βρίσκει σύμφωνος μια τέτοια πολιτικοποίηση. Και αν θέλετε να εθελοτυπείτε σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ψευδοσχέδιο του Επιτρόπου Χόγκαν, γιατί όλοι ήμασταν παρόντες στην παρουσίαση του σχεδίου Τάκτο ανάγκη του κυρίου Χόγκαν που κατόπιν εορτής πολύ καθυστερημένα μας υπέβαλε αυτό το σχέδιο που δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα και την κρίση στην Γεωργία. Και αν θέλετε να αποφύγετε το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σήμερα υπεύθυνη για τη γεωργική κρίση. Κάθε χώρα και φυσικά στηρίζει τη δική της, την εθνική της γεωρική πολιτική και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές πραγματικότητες από τη μία χώρα στην άλλη και όταν ζητούμε μερικές φορές ευρωπαϊκά μέτρα και δεν είναι τα κράτη-μέλη που στυλιτεύουν αυτή την κατάσταση αλλά δυστυχώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπως είδαμε για το γάλα είναι μια πολιτική που σε τελική ανάλυση στερεί από τα κράτη μέλη τον έλεγχο της γεωργίας τους και τα υποχρεώνει να υπαχθούν στην υπεροχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μακάρι να μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και μια συνένεση και να δούμε τι αδυναμίε και τα αρνητικά σημεία τη ε, γεωργική πολιτική του 2014. Γιατί σήμερα, μια διετία μετά, βρισκόμαστε μπροστά σε μια δίρυτη πραγματικότητα. Τι θα κάνουμε, θα στερήσουμε από τα κράτη-μέλη τον έλεγχο τη γεωργία ή θα αφήσουμε τον κύριο Χόγκαν, τον επίτροπο Χόγκαν, να μπορεί ελεύθερα να ελέγχει και να κατευθύνει το έργο της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σαταμπάη. Η κυρία Πετήρ μάθησε μία ερώτηση για τη μείωση από 20% σε 5% του συντελεστή ΦΠΑ για το χείριο κρέας και τα μισά σφάγια θα εφαρμοστεί από την 1η Πρώτου του επόμενου έτους και θα ισχύσει για το γάλα, τα πουλερικά και τα αυγά και μάλιστα όχι προσωρινά, αλλά μόνιμα. Μείωση ΦΠΑ, συντελεστή ΦΠΑ από 20% σε 5%. Περάσαμε αρχικά από από σε 27, 25 και 20% σε 5% στον γαλακτοκομικό τομέα. Το θέμα είναι ποιε θα είναι οι συνέπειε αυτή τη μείωση. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και προτείνω να ξαναδώσουμε το λόγο στους ειδικού, δίνοντάς τους ε, κάποια λεπτά στον καθένα, μερικά λεπτά στον καθένα για να δώσει απαντήσεις. Κύριο κυριος Λέντπερ, παρακαλώ, πρώτος. Τρία-τέσσερα λεπτά για τις απαντήσεις σας. Από εκεί που είσαστε δεν χρειάζεται να σκοθείτε. Ε, ευχαριστώ πολύ. για μια από τις ερωτήσεις που ίσως τέθηκαν για το δικό μου το επιχείρημα ότι η διαφορετική ευελιξία και τις διαφορετικές απαιτήσει τελικά από τα κράτη-μέλη. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Απλώς διαπίστωνα τι συμβαίνει. Εάν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό που συμβαίνει, η δική μου πρόταση είναι να έχουμε περισσότερη διαφάνεια για να έχουν στα χέρια τους οι γεωργοί ένα εργαλείο να μειώσουν μόνοι τους τις διαφορές μεταξύ των κρατών έχοντας περισσότερη γνώση για το πώς οι κανόνες ε, εφαρμόζονται στα άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί από την πλευρά της διοίκησης των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα διευκολυνθεί η διάθεση αυτή που έχουμε για αλλαγή. Από τη δική μας την πείρα είδαμε ότι οι πληροφορίες από άλλα κράτη-μέλη βοήθησαν, βοήθησαν για να αλλάξουμε το πώς γίνονται μερικά πράγματα στη Δανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Σαββατκάι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό απάντησε ο συνάδελφος στην ερώτηση της κυρίας Πέτυρ. Από 1η Ιανουαρίου του 2016 η Ουγγρική κυβέρνηση μείωσε από το 27% στο 5% του ΦΠΑ. Και αναμένεται η σταθεροποίηση ως εκ τούτου της αγοράς χείριου κρέατος τα δεδομένα τα σχετικά με τη φτώχεια που τα παρέθεσα, διότι το χαμηλά εισοδήματα έχουν συνέπεια και στην κατανάλωση χειρίου κρέατος. Και έτσι πιστεύουμε ότι εάν υπάρξει με τη μείωση του ΦΠΑ θα έχουμε ενίσχυση της κατανάλωσης. Για το γάλα πιστεύουμε ότι αντίστοιχα θα πρέπει να εισαχθεί η μείωση του ΦΠΑ όπως και για, το, ε, για τα πουλερικά και τα αυγά. Πιστεύουμε λοιπόν θα πρέπει να πέσει και, και ο ΦΠΑ κατά 5%. Πάντως πρέπει να σημειώσω ότι το, τα κύρια προϊόντα σε χείριο κρέας, όπου έχουμε μείωση του ΦΠΑ, το, το ίμιση Φαγίου, δηλαδή, είναι πιο φτηνά. Έρχονται πιο φτηνά στην αγορά. Και για να απαντήσω σε μια άλλη ερώτηση που ακούστηκε, Η μείωση του φόρου προσθέμενης αξίας θα βοηθήσει, πιστεύω, στην ενίσχυση της κατανάλωσης για τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας, τουλάχιστον στην Ουγγαρία. Αναμένεται ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση κυρίου κρέατος. Τα μέτρα που εισήχθησαν κοστίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό πιστεύω ανεκτό για την οικονομία, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στον προπολογισμό, αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει και να υπολογιστεί κάπου αλλού το ποσό αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σμάτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικές ερωτήσεις απευθύνθηκαν απευθεία σε μένα. Η ερώτηση για, για το κοινωνικό ντάμπινγκ, για παράδειγμα. Σίγουρα θα πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε. Και υπάρχει και το θέμα της έλλειψης κατώτατου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η απουσία τέτοιου ενιαίου κατώτατου μισθού δημιουργεί συνθήκες άνεσου ανταγωνισμού. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα και στην οργάνωσή μας ε, και στο Συμβούλιο Υπουργών. Θα ήταν χρήσιμος ένας κοινό ε, κατώτατος μισθός. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Χέιτεμα για τα 500 εκατομμύρια ευρώ, όλοι γνωρίζουν ότι τα χρήματα αυτά δεν θα εξέλθουν από το αποθεματικό της κρίσης, αλλά από τις άμεσες ενισχύσεις. Αυτό είναι λάθος όμως, το χειρότερο δυνατό. Γιατί θα είναι ελάχιστη η επίδραση στην αγορά. Δεν είναι σωστό αυτό. Το καλύτερο θα ήταν να δοθούν κίνητρα και παρατρήσεις για εξαγωγές σε εμπορικές εκθέσεις, για παράδειγμα. Και πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, θα πρέπει να ξαναπάει ε, στη Ρωσία. Θα πρέπει να έχει απευθείας συνομιλίες με τους Ρώσους. Γιατί είναι πολύ κακό για τους γεωργούς και για τους καλλιεργητές οποροκυπευτικών αυτό το ρωσικό εμπάργο. Και οι ίδιοι Ρώσοι έχουν επηρεαστεί από την πολιτική που εφάρμοσαν και τον εμπορικό του αποκλεισμό. Και 15% του εισοδήματό του οι Ρώσοι το αφιερώνουν στη διατροφή τους. Και τους κοστίζει που δεν έχουν πια την ευκαιρία να απολαύσουν ευρωπαϊκά μήλα ή να μαγειρεύσουν καρμπονάντ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει διαφορετική λύση από τα 500 εκατομμύρια. Βέβαια, όταν προβλέφθηκε το μέτρο, μας χαροποίησε. Αλλά είχαμε πρόβλημα στο ρυθμό εκταμίευσης, που ήταν πολύ αργός. Και ούτε ισότιμα έγινε κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα, ο γαλακτοκομικός τομέας στις κάτω χώρες έκανε κάποιο διάβημα στο Υπουργείο, αλλά ακόμη τα χρήματα αυτά δεν έφτασαν στις τσέπες των Γεωργών. Αλλά χρησιμοποιήθηκε για τον εξυγχρονισμό του κλάδου, στις κάτω χώρες τουλάχιστον. Οπότε η μεμονωμένη γεωργοί δεν είδαν τη διαφορά από αυτό το επιπλέον ποσό. Επίσης, αν δεν υπάρχει εθνικό πρόγραμμα, μένουν αβοήθητοι οι γεωργοί και οι κυπουροί. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι και ο καθένας προσαρμόζεται όπως μπορεί. Αλλά φαίνεται ότι η ίδια η γεωρική πολιτική, η κοινή γεωρική πολιτική δεν βρίσκεται στο πυρόβλητο των κρίσεων, ούτε είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει όπως φάνηκε. Τώρα ήδη συζητούμε την ενδιάμεση αναθεώρηση και ίσως ένα 10% δοθεί για άλλους σκοπούς. Ούτε και αυτό είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό. Πάντως, αν βρεθούν χρήματα και αν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ίσως η διάμεση αναθεώρηση είναι μια καλή ευκαιρία για να δοθούν κίνητρα για τις εξαγωγές. Αυτή είναι η σωστή λύση. Περισσότερες εξαγωγές. Αλλά δεν έχω και μεγάλη αισιοδοξία για την ενδιάμεση αναθεώρηση, ιδιαίτερα να αφαιρεθούν κονδύλια από το γεωρικό προπολογισμό. Τέθηκε μια ερώτηση και για το ρωσικό εμπάργο. Η Ρωσία είναι μια πολύ καλή αγορά και θα πρέπει να την ανοίξουμε και πάλι. Ο πρόεδρος Γιούνκερ παρακολουθεί τις εξελίξεις και παρακολούθησε το ποδηλατικό κύκλο γύρω, ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός και ξέρει πόσο σημαντικό είναι το sprint στα τελευταία μέτρα. Ελπίζω λοιπόν να διδαχθεί από την ανάγκη της επιτάχυνσης ο πρόεδρος Γιούγκερ και να δώσει μια γρήγορη όθηση στις συζητήσεις. Θα πρέπει επίση να δούμε τι ε, επιδόσει των κρατών μελών σε θέματα ευζοία, καλή μεταχείριση των ζώων. Εκεί υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Και αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά το σήμα για να εξασφαλιστεί καλύτερη μεταχείριση των ζώων και οι καταναλωτέ δεν έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε για να λάβουν εμπεριστατωμένα την απόφασή τους. Αναφέρθηκε και το Natura 2000 από κάποιον. Φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας, τα ενδιατήματά μας, τα ζώα, τα πτηνά μας, αλλά όχι εις βάρος των γεωργών μας. Και αυτοί χρήζουν προστασίας. Και μερικές φορές η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της γεωργίας και της φύσης του περιβάλλοντος πρέπει να εθετείται με ευελιξία. Για τα μόνιμους βοσκότοπους, για παράδειγμα. Έχουμε ε, και στις περιοχές Natura τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε, μπορούμε να υιοθετήσουμε γεωργία που θα είναι προσανατολισμένη προς το περιβάλλον και φιλοπεριβαλλοντική, αλλά θα πρέπει να είμαστε δογματικοί. Δεν θα πρέπει να φέρουμε αντίπαλους τους γεωργούς με τους περιβαλλοντολόγους. Δεν είναι αντικρώμενα τα συμφέροντά τους. Μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και γεωργίας. Κάποιος ευρωβουλευτής, ο Εντουάρ Φεράου, δεν κάνω λάθος, είπε ότι η καταλληλότερη λύση είναι η εθνική προσέγγιση. Βέβαια, η Γαλλία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα με τις περισσότερες εξαγωγές. Και μία επανεθνικοποίηση θα φέρει σε πολύ δυσάρεστη θέση τους α, α, Γάλλους Γιώργους, ιδιαίτερα μια διάλυση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν κονδύλια για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αλλά καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με κοινοτικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη για τις επιτυχίες. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις. Να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Σρέγερ. Είπε ότι υπήρχαν μεγάλα κόστη, διότι έγιναν επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευζοία των ζώων. Δύο οδηγίες είχαμε. Η μία είχε να κάνει με την προσαρμογή των ε, μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό βεβαίω ε, είχε κάποιε επιπτώσει υπό την έννοια ότι όταν μιλάμε για μεγαλύτερη κλίμακα εκμεταλλεύσεων μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη εθνισμότητα των χείρων, ε, των νεαρών μάλιστα χείρων που μπορεί να πεθάνουν λόγω των έκτακτων μέτρων που κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε από την οπτική γωνία της κοινωνίας, αλλά και της αγοράς και των γεωργών και των καταναλωτών. Και αν μπορούν όλα αυτά να συμφιλειωθούν μεταξύ του, μπορεί να έχουμε την κατάλληλη βάση και να ε, καταφέρουμε το ισότιμο, του ισότιμου κανόνε για όλου του παραγωγού όλων των χωρών. Όμω, πρέπει να αναλυθούν και δυτικέ πρωτοβουλίε για να καλυφθούν όλε οι ανάγκε. Αυτή είναι μία από τι παρατηρήσει που θέλω να κάνω στην ε, Σουηδία ζητείτε, ε, ζητούνται περισσότερες ε, δυνατότητες στέγασης των ζώων και επίσης συνήθως ζητείται άχυρο για την στέγαση των χείρων, στρομνή. Όμως αν κανείς επιβάλλει τον ίδιο καρόνα στην Ισπανία δεν μπορεί να ισχύσει γιατί έχουν διαφορετικές κλιματικές συνθήκες σε δύο χώρες και διαφορετικές ανάγκες στις κατοχώρες. Εάν δούμε τι ε, πρωτοβουλίε για την ιδιωτικοποίηση του νερού, λόγου χάρη, ή τον αριθμό τετραγωνικών μέτρων ε, που διατίθενται στο χώρο στέγασης κάθε, στάβλησης κάθε χείρου, ε, Σίγουρα κάποιοι κανόνες μπορούν να, να προβλέπονται από την νομοθεσία συνολικά, αλλά είναι πολύ αυστηρά. Στην πράξη μπορεί να αποδειχθούν προβληματικοί. Δηλαδή πρέπει κανείς να θέτει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στην νομοθεσία, αλλά να μπορεί κανείς να το προσαρμόσει. Αλλάξαμε λοιπόν τις διατάξεις, έτσι ώστε να υπάρχει το απαραίτητο περιθώριο για τον ιδιωτικό τομέα και όλα αυτά βάσει των νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε για τις ευρωερωταπαντήσεις σας. Ε, ευχαριστούμε για όλη αυτή τη συζήτηση. Βρίσκω ότι είναι κέρια σημασία για το μέλλον τη όλη συζήτησή μα και του κοινή μα εξέταση του θέματο. Δεν είναι περιττός αυτός ο διάλογος. Ελπίζω ότι ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας. Και σας ευχαριστούμε και εσάς για το φως που ρίξατε στους δικούς μας προβληματισμούς και στα ερωτήματα που θέτουμε εμείς στους ΔΕ. Ολοκληρώνουμε την ακρόαση αυτή στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής μας και περνάμε στο επόμενο μέρος που έχει να κάνει με τον διάλογο, με την ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικέ πράξει για τα θέματα των γεωργικών κρίσεων. Ο κύριο Κορτέ θα έρθει όπου να είναι. Θα σα έλεγα να κάνουμε ένα διάλειμμα για λίγα λεπτά μέχρι να έρθει κοντά μα και να υποφεληθώ αυτών των λίγων, των λίγων δευτερολέπτων για να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Πίτερ Γιάρ. Χρόνια του πολλά, με λίγες μέρε καθυστέρηση. Είναι εδώ στην αίθουσα μαζί μα Να ζήσει. Χθε ήταν τα γενέθλιά σου. Σε χαιρετούμε. Τέσσερα λεπτά τεχνική δια... μέχρι να έρθει εδώ ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ήρθε ο ομιλητής μας. Παρακαλώ λοιπόν να συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όμως πρέπει να καθίστε στις θέσεις σας. Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας και έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων τώρα, όπως γνωρίζετε, με την Επιτροπή για τις Κατεξοδότηση και Εκτελεστικές Πράξεις που σχετίζονται με την γεωργική κρίση. Ευχαριστώ τον κύριο Κόρτα που είναι εδώ θα μας μιλήσει λοιπόν με τις κατεξουδότησες και εκτελεστικές ε, πράξεις που σχετίζονται με την κρίση. Όπως γνωρίζετε, ο Επίτροπος Χόγκαν είχε ανακοινώσει τέτοια μέτρα στο τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας και Ελίας στις 14 Μαρτίου. Μέχρι τώρα έχουμε λάβει μία μόνο κατεξουδότηση πράξη που αφορά το γαλακτοκομικό τομέα, που ε, ε, που ενεκρίθη με την κατεπίγουσα διαδικασία, άρα είναι ήδη ενισχύ Ξέρετε όμω ότι το Κοινοβούλιο έχει ακόμη τη δυνατότητα να διατυπώσει αντιρρήσει. Πρόκειται για μία πράξη σχετική με, την, ε, με το αντίστοιχο νομοθέτημα που απορρέει από τον εκτελεστικό κανονισμό τη ε, Επιτροπής του 2016 για τι συμφωνίες και αποφάσεις στο σχεδιασμό της παραγωγής στο γάλα και τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Καλό λοιπόν τον κύριο Κόρτε να εξηγήσει τους λόγους τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε αυτά τα δύο νομοθετήματα, στις πράξεις, και να μας εξηγήσει και το περιεχόμενο πιθανών άλλων ε, σχεδίων πράξεων, εκτελεστικών ή κατεξουσιοδότηση που μπορεί να σχετίζονται με τη γεωργία και την γεωργική κρίση πάνω απ' όλα και ενδεχομένω είναι υπό επεξεργασία σε επίπεδο Επιτροπής και γενική διεύθυνση Γεωργία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Οντριέ. Και στο συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Κατά την άφηξη, σας ευχαριστώ πολύ που προβλέψατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την κατάσταση στη Γεωργία. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητική κατάσταση στο γεωργικό τομέα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και κυρίως στο γαλακτοκομικό τομέα, στον τομέα του χείριου κρέατος και γι' αυτό είναι απολύτω απαραίτητο να γίνει σημερινή αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας δώσω ενημέρωση για τις ε, επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις πράξεις που εισήγαγε από την τοποθέτηση ενώπιον της Ολμέλης του Κοινοβουλίου του Επιτρόπου Χόγκαν πριν από δύο εβδομάδες. Στα αγγλικά τώρα δεν σκοπεύω κύριε Πρόεδρε να επισέλθω στη λεπτομέρεια του κάθε μέτρου που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Μάρτιο, όπως ξέρετε, ο Επίτροπος Χόγκαν προεξήγηλε 13 διαφορετικά πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης στο γεωργικό τομέα. Σύμφωνα όμως και με το έτοιμά σας, θα εστιαστώ στις κατεξουσιδότητες πράξεις σήμερα. Βεβαίω υπάρχει έργο να εξελίξει. Ε, είμαστε στη φάση ε, διαχείρισης των ε, μέτρων ιδιωτικής αποθήκευσης Επίσης έχετε καλέσει εσείς τον κύριο Βέμαν και τον, τον πρόεδρο αλλά και άλλους, τον κύριο Μωρό και άλλους, ε, να σας ε, δώσουν πληροφορίες και ε, μάλιστα έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα κονδύλια για την προαγωγή των γεωργικών προϊόντων. 13 εκατομμύρια θα θυμάστε είχαν διατεθεί για το γάλα, για τη Συρία θα διατίθεται. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα γάλακτος που θα διατίθεται προς πόσιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης ε, αναζητούμε νέες διεξόδους αγοράς. Ε, Επισκεφθήκαμε την Ιαπωνία και την Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα ακριβώς για το, μέσα στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων αγορών τώρα για να ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις από την ομιλία του Επιτρόπου ενώπιον σας πριν από δύο εβδομάδες. Το πρώτο μέτρο δεν απαιτεί συμφωνία του Κοινοβουλίου. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Έχει να κάνει με την αύξηση του ανωτάτου ορίου παρέμβασης αποκορυφωμένης ε, σκόνης γάλακτος. Έχουμε 109.000 τόνους κατά μέγιστον και 50.000 για το βούτυρο 100.000 για, για την αποκορυφωμένη σκόνη γάλακτο και αντίστοιχα για το βούτυρο 50.000. Και πέραν αυτών, α, των αντατονορίων, πρέπει να προχωρήσει σε πληστηριασμό... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν δεν είμαστε πια στη σταθερή τιμή, αλλά στο σύστημα των πληστηριασμών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό των άμετων αυτών 218 δηλαδή χιλιάδε τόνου για την αποκορυφωμένη σκόνη γάλακτο και 100.000 για το βούτυρο. Απόφαση που ταχύτατα ενέκρινε και το Συμβούλιο και έτσι έχουμε τώρα τη δυνατότητα να εξακολουθήσουμε να παρεμβαίνουμε στην σκόνη και το βούτυρο για πολύ μακρύτερο διάστημα μέχρι να φτάσουμε στα ε, αργοτόρια, αντίστοιχα του 200, των 218.000, όπως είπα, για την αποκορυφωμένη σκόνη παραπτώση. Το γεγονό βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει πολύ μεγάλες ποσότητες δεν είναι καλό δείγμα. Δείχνει δηλαδή ότι η, Ευρωπαϊκή, ότι η αγορά δεν απορροφά την σκόνη γάλακτος. Για το βούτυρο πρόβλημα δεν υπάρχει. μόνο υποκορυφωμένη του κόνη γάλακτος ε, για να ανησυχίε και αυτό δείχνει ότι η κρίση στην αγορά γάλακτος είναι βαθιά. Αυτό λοιπόν έχει προχωρήσει. Από την προηγούμενη εβδομάδα ισχύουν ε, τα νέα ανώτατα όρια. Στο γαλακτοκομικό τομέα πάντα, κύριε Πρόεδρε, το επισημάνω τέλος του κι εσείς, έχουμε δύο μέτρα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενθαρρύνει της εκούσιες συμφωνίες μεταξύ κτηνοτρόφων προκειμένου να σχεδιάσουν καλύτερα την ε, παραγωγή γάλακτος. Ε, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υπό το 222 της ε, αγορά, το άρθρο λέει, της κοινής αγοράς, συνθήκης κατά εξουσιοδότηση πράξη, αλλά και εφαρμοστική πράξη, που έχουν υιοθετηθεί και βρίσκονται ενισχύ από τις 13 Απριλίου και θα ισχύσουν για 6 μήνες έως τις 12 Οκτωβρίου του 2016 συγκεκριμένα. Η κοινή οργάνωση αγοράς, βασικός κανονισμός εν προκειμένου, επιτρέπει παράταση για άλλους 6 μήνες κατά μέγιστο των μέτρων. Άρα η περίοδος μέσα στην οποία μπορούν να συναυθούν αυτές οι ακούσεις συμφωνίες ε, ήδη τρέχει, ήδη είναι ενισχύ. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω πολύ σύντομα γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό το νομοθέτημα και γιατί καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, το υποστηρίξει με τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο της ε, επαλήθευσης της κατεξουσιοδότησης πράξης. Αν κοιτάξουμε τις... Γιατί είναι σημαντικό λοιπόν το μέτρο αυτό. Γιατί πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γαλακτοπαραγωγούς να παράγουν λιγότερο και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το καταφέρουμε αν δεν έχουμε ζητήσει μα αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Για να δούμε λοιπόν την κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τρεις παράγοντες που προξενούν δυσκολίες. Πρώτον, έχουμε μια σοβαρή κάμψη στις παγκόσμιες ε, τιμές, στην παγκόσμια αγορά. Ε, είναι κάτω, είναι πολύ χαμηλά οι τιμές γάλακτος, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλο τον κόσμο. Ε, και αυτό οφείλεται και στις χαμηλές τιμές των βασικών αγαθών που επηρεάζουν όχι μόνο το γάλα αλλά πολλά βασικά αγαθά και της, λόγω της μείωσης της ζήτησης ιδιαίτερα στην Κίνα και αυτά συνιστούν τον πρώτο λόγο. Ο δεύτερος λόγος δυσκολιών για το γαλακτοκομικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς σχετίζεται με το ρωσικό εμπάργο. που ξέρετε αποτελούσε η Ρωσία πολύ σημαντική αγορά για το γαλακτοκομικό τομέα της ε, Ευρώπης. Από τον Αύγουστο του 2014 έχει κλείσει αυτή η αγορά. Τρίτος λόγος είναι η εκπνοή των ποσοστώσεων γάλακτος ε, τον Απρίλιο του 2015 που οδήγησε σε σοβαρή αύξηση της παραγωγής γάλακτος και αυτό βέβαια εντείνει τις δυσκολίες στις αγορές. Λόγω των δύο πρώτων παραγόντων που σας ανέφερα ήδη υπήρχαν δυσκολίες και αυτές εντείνονται. Βλέπουμε δηλαδή στην Ευρώπη αύξηση της παραγωγής γαλάκτος κατά 4 με 5% γενικά στην Ευρώπη σε όλο τον τομέα από την ε, εκπνοή των ποσοστώσεων. Βέβαια οι διαφορές ανά κράτος μέλος είναι σημαντικές. Δεν είναι σε όλα τα κράτη-μέλη ε, τόσο υψηλή η αύξηση, αλλά η τάση και ο μέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 4 5%. Και αν κοιτάξετε αντίστοιχα τα στοιχεία στην ε, ιστοσελίδα του γαλακτοκομικού τομέα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει αυτή η τάση αυξητική λοιπόν στην παραγωγή. Αυτά είναι τα μέτρα που προσπαθούμε, να, ε, Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να εισαγάγουμε μέτρα προκειμένου να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να οργανωθούν, να οργανωθούν μεταξύ τους μέσα σε οργανώσεις παραγωγών διατομεακά ή διακλαδικά, διεπαγγελματικά όπως λέμε στα γαλλικά, interprofessionnel, μέσα από συνεταιρισμούς, προκειμένου να μπορέσουν οργανωνόμενοι να ε, συμφωνούν από κοινού περί της ε, παραγωγής γάλακτος. Ε, κανονικά θα έπρεπε αυτές ε, οι συνεννοήσεις να απαγορεύονται δυνάμει της νομοθεσίας του ανταγωνισμού γιατί δεν επιτρέπεται παραγωγή να συμφωνούν και να ορίζουν μέσα από μια ε, συμφωνία που θα ισοδυναμούσε με καρτέλ βέβαια ε, τον έλεγχο της παραγωγής. Τώρα με την πρόταση αυτή έχουμε ε, στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς του ή άλλως τη δυνατότητα να εξαιρεθούν οι παραγωγοί εφόσον όμως είναι οργανωμένοι γάλακτος από την απαγόρευση αυτή και σε αυτό το μέτρο ακριβώς προβαίνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα και έτσι προσφέρουμε μια ασπίδα, μάλλον απελευθερώνουμε μια ασπίδα που προσφέρει τόσο άλλο η κυνηγή οργάνωση αγοράς, η πολιτική και επιτρέπει έτσι στον, γεωργό, ε, στον παραγωγό γάλακτος να περιορίσει την παραγωγή του ε, για ένα διάστημα. Πρόκειται για μια νέα διάταξη που εισήχθη το Δεκέμβριο του 2013 με τη δική σας βοήθεια στην κοινή οργάνωση αγοράς για το γάλα και τώρα είναι η πρώτη φορά που δραστηριοποιείται το μέτρο αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ ενώπιον σας σήμερα αλλά και γενικότερο ο Επίτροπος δεν σταματά να απευθύνει εκκλήσεις προς το γαλακτοκομικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και δυνατότητα. Για να συνοψίζω, Πρόεδρε, και ήθελα πολύ σύντομα να εκθέσω κάποιες άλλες σημαντικές ε, παρατηρήσεις, πιστεύω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε κίνηση άλλη μια διαδικασία για ένα παρατηρητήριο αγοράς κρέατος. Ξέρετε ότι λειτουργεί ήδη ένα τέτοιο παρατηρητήριο εδώ και δύο-τρία χρόνια. Ο Επίτροπος Χόγκαν Υπάρχει παρατηρητήριο για το γάλα εδώ και μερικά χρόνια. Ο Επίτροπος Χόγκαν είχε προεξαγγείλει και ένα αντίστοιχο παρατηρητήριο για το κρέα, Ε, πρακτικά μόνο μέσα από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μπορούμε να συστήσουμε ένα τέτοιο παρατηρητήριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία συνίσταται από εκπροσώπους που έχουν ανταποκριθεί σε έναν ε, διαγωνισμό για ειδικού έχει ολοκληρωθεί αυτό ο διαγωνισμός, μπορούν να διατυπωθούν οι αιτήσει μέχρι τις 15 Μαΐου από τους ενδιαφερομένους. Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμό και μπορούν να διατυπωθούν οι αιτήσει. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συσταθεί η αντίστοιχη επιτροπή, το παρατήριο δηλαδή για το κρέα, ε, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τι ελληνέ διακοπέ. Και άρα θα παρακολουθούμε, πιστεύω, εγκύτερα τι εξελίξει και για το ε, χείριο, αλλά και για το βόλιο και το μοσχαρίσιο κρέα. Αυτούς τους τρεις τομείς τα καλύπτει δηλαδή, το παρατηρητήριο για τα οπορικά και λαχανικά. Οι στατιστικές των συναλλαγών, οι εμπορικές στατιστικές και τα δεδομένα που έχουμε δείχνουν και είναι αυτό καθησυχαστικό ότι έχουν μπορέσει περισσότεροι παραγωγοί να προσαρμοστούν στην απώλεια της ρωσικής αγοράς λόγω του εμπάργου. Έχουν βρει εναλλακτικέ ε, διεξόδους για τα προϊόντα τους. Ξέρετε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2014 παρενέβη με συγκεκριμένα μέτρα αμέσως για να προστατεύσει τον τομέα των απορρολαχανικών καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτα ε, προϊόντα προϊόντα με πολύ μικρή διάρκεια ζωής, ένα εκατομμύριο τόνοι όπορο λαχανικών έχουν αποσυρθεί από την αγορά με συνολικό κόστος των μέτρων αυτών τα τελευταία δύο χρόνια 262 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο που παραμένει ενισχύει προς το παρόν εκπνέει στα τέλη Ιουνίου και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει νέο μέτρο, κάτω εξουσιοδότηση πράξη, εν προκειμένου, δεύτερη κατεξουδότηση πράξη κύριε Άντριε, που θα δείτε σύντομα, με την οποία θα παρατηρείται για ακόμη ένα χρόνο το εφιστάμενο πρόγραμμα. Δηλαδή θα πάει μέχρι, την πρώτη, μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2017, εκτός και αν μέχρι τότε έχει ε, αρθεί το εμπάρκο. Πράγμα το οποίο θα ήταν καταπληκτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινάμε με δεδομένη την παράταση για ένα χρόνο του μέτρου. Με μεγάλη προσοχή μελετούμε την ανάγκη να προσαρμοστεί το εφιστάμενο σύστημα. Και μια και πρόκειται για το τρίτο έτος λειτουργίας του συστήματος και δεδομένου ότι έχουν βρει πολλοί, όπως είπα από τον τομέα, εναλλακτικέ διεξόδους, ο προϋπολογισμός που σχεδιάζουμε να δώσουμε στο σύστημα αυτό ε, θα είναι πολύ ε, περιορισμένος, όπως περιορισμένες θα και οι ποσότητες. Θα έχουμε λοιπόν μία πρόταση συγκεκριμένου ποσού στο σύνολο και ποσοτήτων ανακράτος μέλος σε σχέση με την κατάσταση του 2014 και αυτό, με αυτό που βλέπουμε σήμερα, κοιτώντας τα μέτρα και ρωτώντα ε, του ρωτώντας τους ειδικού μου τι, με τι πρόβλεψη είχαν ξεκινήσει τα μέτρα που εκπνέουν τώρα, τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή από τη στιγμή που εισήξαν τον Ιούνιο του 2015, 35% μόνο των μέτρων αυτών αξιοποιήθηκαν, 35% το οποίο δείχνει βέβαια ότι υπήρχε λιγότερη ανάγκη για τα μέτρα αυτά και γι' αυτό ακριβώς θα είναι πιο περιορισμένος ο όγκος στην πρόταση αυτή κατεξουδότηση πράξης. Και η χρηματοδότηση εν τέλει. Ο Επίτροπος έχει καταστήσει, νομίζω και ενώπιον της Ολομελίας, σαφές ότι αυτή τη στιγμή ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν επιτρέπει χρηματοδότηση για να υποστηριχθούν οι παραγωγοί που θα ήθελαν να μειώσουν την παραγωγή γάλακτος. Αλλά συζητήσαμε και ανοίξαμε τη δυνατότητα, εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα ουσιαστικά για τα κράτη-μέλη να προσφέρουν κρατικές ενισχύσεις, στηρίζοντας τους παραγωγούς που βρίσκονται σε δυσκολία, πέραν των υφισταμένων ενισχύσεων και έχουμε ε, απευθύνει τις σχετικές εγκυκλίου στα κράτη-μέλη μέχρι 15.000 ευρώ ανά παραγωγό κατέτος για τους τομείς που βρίσκονται σε κρίση, σε δυσκολία επιτρέπεται να διαθέσουν επιπλέον τα κράτη. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ε, ένα πρόσθετο στοιχείο, ότι αυτές οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να πάρουν τη μορφή δανείων, που βέβαια θα επιστρέφουν ή εγγυήσεων και αν στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης δεσμευτεί ο παραγωγός ή να μειώσει έστω να σταθεροποιήσει την παραγωγή του, μπορεί να πάρει και τη μορφή καθαρής ενίσχυσης αυτή η υποστήριξη και άρα δεν θα χρειάζεται να αποπληρωθεί. Όμως μόνο εφόσον από πλευράς του παραγωγού αναλαμβάνεται αυτή η δέσμευση. Και εδώ μιλούμε και για το γαλακτοκομικό τομέα ιδιαίτερο, δηλαδή να δεσμευθεί ο παραγωγός να παράγει λιγότερο ή τουλάχιστον να μην παράγει περισσότερο γάλα για να ανοίξει το σύστημα κρατικών ενισχύσεων προ τον παραγωγό. Για να μην φτάσουμε δηλαδή κρατικέ ενισχύσει να ε, πηγαίνουν σε παραγωγού οι οποίοι ενισχύουν την, αυξάνουν την παραγωγή του και να χρηματοδοτείται η αύξηση τη παραγωγή. Με αυτά τα μέτρα νομίζω. Σας έχω ε, συμπληρώσει την εικόνα από τα όσα έχει πει και ο Επίτροπος Αναπλών Ολομέλειας πριν από δύο εβδομάδες για τα μέτρα της Επιτροπής. Ελπίζω σύντομα να μπορέσετε να δώσετε και εσείς το πράσινο φως στην κατεξουδότηση πράξη που σας έχει υποβληθεί για τις ε, εκούσες συμφωνίες περί, περιορισμού της παραγωγής και του συνεταιρισμού για το γάλα και ελπίζω αργότερα να έρθει και η ώρα για τα όπορο λαχανικά που θα ε, ακολουθήσουν σε μια-δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ξεκινά, συνάδελφοι. Παρακαλώ, κύριος Δάντα, Πρώτος, γιατί είναι και εισηγητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι πληροφορίε που μας έδωσε ο κύριος Κόρτε δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπήκε σε φάση διαχείρισης ε, της κρίσης από ψυχολογική άποψη. Από ψυχολογική σίγουρα, αλλά και από ηλική δεν είμαι βέβαιος από ουσιαστική άποψη. Γιατί δεν πιστεύω ότι όλοι οι επίτροποι και δύο αρμόδιες Επίτροπες προϋπολογισμού είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη κατάσταση των Ευρωπαίων Γεωργών. Έκανα ένα μικρό υπολογισμό και η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να δοθεί από τα κράτη-μέλη είναι 15.000 ευρώ το χρόνο. Και σήμερα σε πολλές χώρες η παραγωγή μας λένε ότι χονδρικά η τιμή πώληση δεν καλύπτει καν το, το κόστος. Και έχει απώλεια, έχουν απώλεια τους 8 με 10 λεπτά. Οπότε για κάποιον παράγει 150.000 ε, λίτρα το χρόνο, ε, τα 15.000 ε, δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν να περισσώσει τις απώλειες και τις ζημίες που έχει υποστεί ούτε ο περιορισμός της ε, εθνικές ενισχύσεις ε, είναι ε, σωστή λύση κατά τη γνώμη μου. Γιατί έχουμε κοινή γεωργική πολιτική και αν σε κάθε κρίση επιρρύπτουμε τις ευθύνες στα κράτη-μέλη, τους αφήνουμε να, βγάλουμε, να βγάλουν μόνο τους τα σπασμένα, να πληρώσουν μόνο τους τα σπασμένα, τότε προς τι κοινή πολιτική. Νομίζω λοιπόν πέραν του αρμοδίου επιτρόπου Γεωργίας θα πρέπει να προσφύγουμε στο σύνολο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο. Δεδομένων των ε, κατεξουδότηση πράξεων που μας προτείνονται, νομίζω ότι το μόνο μέτρο, μέτρο που μπορεί να μας βοηθήσει για την κρίση είναι να εθαρρύνουμε γενικώ τους παραγωγούς στην Ευρώπη να περιορίσουν όλοι λίγο την παραγωγή τους. 2 ή 2,5% υπέρβαση της ε, προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση αντιστοιχεί ε, σε ένα ρυθμιστικό παράγοντα που κυρίως προέρχεται από το, τις ζωοτροφές. Καλύτερα λοιπόν να έχουμε βοήθεια για την μείωση παραγωγής παρά να πρέπει ε, να αποθεματοποιήσει, να ξαναθέσει ε, σε εμπορία αργότερα το προϊόν που έχει παράγει, είτε πρόκειται για ένα γάλα σε σκόνη, είτε για βούτυρο. Οπότε θα πρέπει και αυτό το δεχόμενο να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, στην για το πράξη που ε, πε, επεκτείνει στους ελευθερισμούς στο σύνολο των μέτρων, πιστεύω ότι αυτή θα την υποστηρίξουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τα χρηματοοικονομικά μέτρα που θα συνοδεύσουν το μέτρο. Σε ό,τι αφορά τα απορροκυπευτικά, η ανάλυση των αγορών δείχνει ότι σε μερικές χώρες βρέθηκαν διέξοδοι και αλλού από ότι στις παραδοσιακές διάβλους. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η προσπάθεια ανέβρεσης νέων αγορών και νέων διεξόδων. Αλλά μόλις τώρα μπαίνουμε ε, σε ουσιαστική περίοδο παραγωγής οποροκυπευτικών. Και τον επόμενο 1,5 μήνα θα διαμορφώσουμε πληρέστερη εικόνα για την αγορά οποροκυπευτικών. Οπότε μόλις λάβουμε την κατεξότηση πράξη θα την συγκρίνουμε με την πραγματικότητα στην αγορά, γιατί θα ξεκινήσει παντού η παραγωγή στην Ευρώπη και θα φτάσει στο αποκορύφωμά της ε, στις επόμενες εβδομάδες ε, για τα απορροκυπευτικά. Σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις, διευκρινήσεις και τις ε, ιδέες σας. Η κυρία Μίλλορ έχει το λόγο. Κύριε Κόρτε, κύριε Κόρτε, κύριε Κόρτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, για τα όσα μας είπατε. Βλέπω βεβαίως ε, στη Γερμανία ότι δεν θέλουν συνεννοήσεις ε, οι γαλακτοπαραγωγοί, συνεταιρισμούς έχουν τους ή άλλους. Εγώ γνωρίζω κάποιον ο οποίος φαίνεται να έχει ακούσει ότι θα πρέπει να μάλλον να υποστηρίζει ένας από τους ε, γαλακτοπαραγωγούς ενός συνεταιρισμού ε, να υποστηρίζει την ιδέα της μείωσης της παραγωγής. Όλοι οι άλλοι όμως βλέπουν ότι υπάρχουν τόσο αυστηρά κριτήρια τα οποία δεν τους επιτρέπουν και τις κινήσεις. Θέλουν περισσότερο να διατηρηθούν στα ύψη τους οι τιμές και γι' αυτό πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να βρούμε λύσεις διαφορετικές όπως και ο κύριος Δες. Πιστεύω ότι Πρέπει να ξαναμελετήσουμε τις προτάσεις για τη διάθεση στην αγορά γάλακτος για παγωτό, για άλλες χρήσεις στην παραγωγή, στη μεταπίεση, για βούτυρο ενδεχομένως και αυτά τα 15.000 ευρώ σε ενίσχυση στη Γερμανία Ήδη έχει δοθεί σχετική υπόσχεση από το, δήλωση μάλλον από τους αρμόδιους για τα γεωργικά υπουργούς. Δεν θέλουν να διαθέσουν τα ποσά αυτά. Προς το παρόν δεν προχωρούμε περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη ξανασδρίχνουν τον μπαλάκι προς την Κομισιόν. Δεν ξέρουμε αν θα σταματήσει αυτό το πινκ-πονγκ γιατί νέο χρήμα δεν υπάρχει και διαρωτώμε εάν υπάρχει δυνατότητα σε επίπεδο ευρωπαϊκό να ε, αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις. Και στην Ολομέλεια, όπως το είπα, εγώ νομίζω ότι μια πρημοδότηση για τον περιορισμό των του ζωικού κεφαλαίου αλακτοφόρων αγελάδων θα ήταν χρήσιμος λύση. Το έχω πει στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ένα μέτρο δηλαδή επιδότηση σε μια πριμοδότηση για προσαρμογή στην αγορά και μόνο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των ποσοτήτων γάλακτος που εισραίουν στην αγορά. Ευχαριστούμε κύριε Σχόισλινγκ. Πρόεδρε. Κυρία Μίλλερ, να, μας μιλάτε δηλαδή για πρημοδότηση φαγής, άρα γυρνάμε πίσω στη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία του 60 που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ε, σφάζουμε τις αγελάδες γιατί φορετικά αυξάνονται τα αποθέματα γάλακτος. Μα δεν μα έχει εξηγήσει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση τώρα από τι συζητήσει που έχουμε κάνει για το γεγονό ότι ο Επίτροπο δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει. Μπορεί να μην συμφωνούσαμε σε όλα τα ζητήματα, βέβαια, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να μειωθούν ε, οι ποσότητε του γάλακτο. Τώρα μα λέει η Επιτροπή, Α, τα κράτη-μέλη πρέπει να το πράξουν αυτό. Μα τι να σα πω, ότι, και, ότι προγράμματα και να προτείνουν τα κράτη-μέλη και να πούνε να συνεταιρισμοί κτλ. Να, να τα βρούνε με το γαλακτοκομείο κτλ χρειάζεται ένα μέτρο ενιαίο για την Ευρώπη. Ένα μέτρο το οποίο θα φέρει αποτελέσματα. Δεν μπορεί να μειώσει ο ένας γαλακτοπαραγωγός και οι άλλοι να συνεχίζουν να παράγουν τις ποσότητες που είχαν και στο παρελθόν. Ευρωπαϊκό μέτρο χρειάζεται. Μέτρο το οποίο θα ε, επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη σε θέση να χρηματοδοτήσουν τον περιορισμό των ποσοτήτων γάλακτος στο εσωτερικό τους. Δεν έχουμε μπορέσει λοιπόν να βρούμε καμία λύση σε αυτή την ευρωπαϊκή κρίση. Λέτε ότι θα έχετε ένα παρατηρητήριο τώρα και για το κρέας. Μα τι θα παρατηρήσει το παρατηρητήριο, ότι είναι κακές, κακά τα επίπεδα των τιμών. Χαίρομαι πολύ. Έχετε τίποτα να προτείνετε. Μετά χρειάζεται να υπάρχουν εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν ε, να πούμε εάν η κατάσταση είναι αυτή, κατευθύνουμε την αγορά προς τα εκεί, προς τα ε, εδώ. Χρειάζεται κάποια κατεύθυνση, καθοδήγηση για την παραγωγή, για την αγορά. Όσο δεν γίνεται αυτή η συζήτηση, πώς θα καθοδηγήσουμε την παραγωγή, κάθε συζήτηση είναι περίτη. Τι θα το κάνουμε, θα, θα, πλη, θα πλημμυρίσουμε τα κράτη σε σκόνη αποκοροφωμένη γάλακτος ή σε βούτυρο. Δεν υπάρχουν σοβαρές λύσεις. Τι θα πάμε, μας λέει ο πίτροπος... Ε, υπάγεται ανά των κόσμων και πωλείται το γάλα. Πολύ καλά να το κάνουμε, αλλά δεν γίνεται. Στην πράξη δεν φέρει αποτέλεσμα. Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκές λύσεις με ευρωπαϊκά μέσα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να σωθεί ο τομέας. Θα έχουμε όλο και μεγαλύτερες κρίσεις. Ήδη βλέπουμε γάλακτοπαραγωγούς με τιμές πώλησης κάτω από τα 20 λεπτά του ευρώ. Μιλούμε για μεγάλη οικονομική κρίση. Μιλούμε για καταστροφή ολόκληρου τομέα παραγωγής. Τι θα κάνει επιτέλους η Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λουβαζό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τι γεωργικέ κρίσει και τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τι αντιμετωπίσει, ασθένοντα θα έλεγα, δεν καταφέρνετε τίποτα. Μια πρόσφατη μελέτη για την κατάσταση τη γαλλική γεωργία που βρίσκω ότι είναι πολύ καλή, κάνει μια καλή επισκόπηση της κατάστασης. 53% των γεωργών στη Γαλλία αυτή τη στιγμή ε, έχουν μείωση των εισοδημάτων τους και 14% από αυτούς, 14%, πιστεύουν ότι καλό θα ήταν να εγκαταλείψουν την δραστηριότητά του ήδη φέτο. Δραματικό, γιατί διότι ακριβώ του έχει πλήξει η μείωση των εισοδημάτων και το δυσβάσταχτο γραφειοκρατικό άχθο. Ο Επίτροπο Χόγκαν εδώ έχει υποστηρίξει την απελευθέρωση των ποσοστών γάλακτο και προκάλεσε την κρίση του χείριου και του βόλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είδα και με τα προκυπευτικά, μια σοβαρότατη κρίση, η οποία συνδέεται με την κρίση των δημετριακών. Επίση σημαντική. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι έχουν κοστό παραγωγής και το ξέρετε όλοι πολύ ανώτερο από, το, από την τιμή πώληση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ΚΑΠ. Και πράγματι αυτέ είναι οι Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά στήρε συζητήσει. Έκτακτα μέτρα χρειάζονται για να επιληθεί η κρίση, αλλά δεν έχουν αναλυθεί. Θα έπρεπε να υπάρχει ριζοσπαστική αλλαγή στην κοινή αγροτική πολιτική τη Ευρώπη, που θα έπρεπε να ξαναδώσει όλε τι δυνατότητε στα κράτη-μέλη για να αναλάβουν την εθνική του κυριαρχία, να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών γεωργιών και να μπορέσουν να χτυπήσουν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι οι κλειδονισμοί τη γραφειοκρατία που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί και που προκαλούν και υπερφόρτωση και άγχος. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια πολιτική που δεν θα οδηγεί συνδυαστικά προ τα κάτω τι τιμέ, που δεν θα ωφελεί μόνο τι μεγάλε βιομηχανίε πλήττοντα του μικρογεωργού. Και πιστεύω ότι αυτέ τι ιδέε πρέπει να εξετάσει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι το γεωργικό μα μοντέλο πρέπει να ξανασχεδιαστεί. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα τη γεωργία για να βασιστούμε στο αμερικανικό μοντέλο, μια υπεργεωργία που θα αντιμετωπίσει μόνο τον ανταγωνισμό στι διεθνεί αγορέ, ή μια γεωργία παραδοσιακή, ξανακατοικ ανακτώντας την εσωτερική μας αγορά και ανακτώντας την επισητιστική μας κυριαρχία. Εδώ η ευρωπαϊκή πολιτική και πάλι είναι αντιφατική, είναι άσυνεπής, είναι κάτι που μας αφήνει άφωνος και βλέπω εδώ πολλούς βουλευτές, ε, είναι αρκετοί ήδη σήμερα, που στηρίζουν αυτή τη γεωργία. Καταλαβαίνω όμω ότι έχουν αειδιάσει πια, έχουν ε, απειδήσει οι γεωργοί τη Ευρώπη με την ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι σαφώ αυτή ε, αυτή η κατάσταση. Και ο λόγο είναι ότι περισσότεροι από του ερετούς εδώ δεν είναι γεωργοί. Δεν του αφορά άμεσα το θέμα καν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μποβέ. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι αυτά που είπε ο κύριος Νταντά ε, είναι λογικά. Και με το δικό του τον τρόπο βρήκατε ήταν σαφέστατος έδειξε πόσο διαφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι πραγματικά υπάρχει φοβερή ασυνέπεια στις πολιτικές που προτείνονται και η ασυνέπεια αυτή δεν θα επιτρέψει να επιληθεί κανένα πρόβλημα. Επαναθνικοποίηση των βοηθειών. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη να υποκαταστήσουν την ευρωπαϊκή, επιτοπή, ε, την ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό καταφέραμε με τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική και βλέπουμε που φτάσαμε σήμερα. Συνολικά λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε πάρει στραβό δρόμο. Είναι πραγματικά συνεπέ να ζητάμε από του γεωργού του ενό ή του άλλου κλάδου να μειώσουν την παραγωγή του, ενώ άλλοι συνεχίζουν να την αυξάνουν. Δηλαδή στι περιπτώσει αυτέ υπάρχει μια διαρκή στάση να αυξάνονται τα προβλήματα, αν δεν υπάρχει μια συνολική πολιτική για να ελέγξουμε τον όγκο παραγωγή, θα οδηγηθούμε σε καταστροφή. Και δεν μιλάω απλώ για το γάλα που είναι μια κλασική περίπτωση, αλλά το ίδιο για τι ονομασίε προέλευση, διότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά αρνήθηκε όταν ε, μελετήσαμε τα, τη δεσμή για το γάλα να ξαναδεί τον όγκο παραγωγή που επιτρέπεται για τι ονομασίε προέλευση με τον έλεγχο των τιμών ταυτόχρονα. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα του γάλα παραγωγικό τομέα. Για τον τομέα παραγωγής κρέατος. Μιλήσατε για κρίση, αλλά δεν θίξατε καν ένα θέμα που είναι κέρια σημασία για τους προσεχείς μήνες και τα προσεχή έτη. Δηλαδή, οι συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αυτή τη στιγμή συνάπτονται με τον Καναδά, οι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ και οι διαπραγματεύσει με, με τη Μερκοσούρ. Σήμερα η εάν αποδεχτούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και την έκβασή τους, 20 και 30, έως 30% ε, του ζωικού κεφαλαίου των βοηδών, του κρέατος, θα αποδιοργανωθούν. Ε, θα το χάσουμε. Δηλαδή η κρίση που θα μας πλήξει θα είναι πραγματικά δραματικών διαστάσεων. Εδώ μιλώ μόνο για τα βοηδή. Εάν προσθέσουμε και τους χείρους, η κατάσταση θα είναι παρόμοια. Ο Καναδάς θα εξάγει χείριο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτοί θα θέλουν ε, να εξάγουν χείριο. Το ίδιο και ο Μερκοσούρ. Οπότε περνάμε πάλι σε μία διόγκωση ε, και μία εκτατική, εκθετική μάλλον ε, διάσταση του προβλήματος. Πρέπει να δούμε λοιπόν όλες αυτές τις, ελευθερίες, όλες αυτές τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Και νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να πούμε καμία συμφωνία. Τέλεια και παύλα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Χόιμπλουχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Μποβέ το είπε μόλις τώρα. Έχουμε να κάνουμε με μια όλο και περισσότερο ασυνάρτητη πολιτική και βεβαίως μπορούμε να χαιρόμαστε για το ότι βλέπουμε από πλευράς του Επιτρόπου συζήτηση για μείωση των ποσοτήτων. Αλλά όταν μιλούμε για εκούσια σχέδια δεν καταλαβαίνουμε πού πάμε. Και πρέπει να το πούμε και θα συμπληρώσω εδώ ότι θα χάσουμε παραγωγή ανά επιφάνεια σε γάλα εάν τώρα δεν αναλάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε τις ποσότητες. Ήδη βλέπουμε την περίπτωση της Ρουμανίας που πλημμύρισε από ευρωπαϊκό γάλα και δεν είναι πλέον σε θέση περιφερειακή και τοπική παραγωγή να διατηρήσουν τη θέση του στην αγορά. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να επισημάνω. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε βεβαίως πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να ε, παραμένουν βιώσιμοι οι κτηνοτρόφοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι νομίζω να επιδοτηθούν. 3,1 δισεκατομμύρια ε, ε, ευρώ σε επιδοτήσεις για το γάλα χάνονται εάν η τιμή του γάλακτος πέφτει όπως βλέπουμε στα 20 λεπτά του ευρώ ανά Ποιο θα τα επιδοτήσει, πώ θα τα δώσει τα χρήματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να μιλούμε λογικά για μέτρα τα οποία θα δώσουν αποτελέσματα. Χρειάζεται υποστήριξη ανά έκταση για ολόκληρη την Ευρώπη και με τρόπο δεσμευτικό. Merci, Ευχαριστώ, κυρία Σρέιρ. Ευχαριστώ. για το θέμα των κονδυλίων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Την περασμένη εβδομάδα είχα επαφές ε, με κτηνοτρόφους και γαλοπτοπαραγωγούς ε, και μου είπαν ότι μακάρι να έπαιρναν απευθεία αυτά τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί γιατί ξέρουν πώς να τα αξιοποιήσουν. Τώρα, η ερώτηση για τις 15.000 ευρώ το χρόνο το πολύ οργό. Μπορεί όμω να έχουμε ένα γεωργό που έχει 20 εκτάρια και άλλο να έχει 2.000 εκτάρια. Ο Πίτερ δεν κάνω λάθος, έχει 20.000 εκτάρια δεδομένης καταγωγή του. Οπότε 15.000 για ένα μικρό καλλιεργητή είναι μάνα εξ ουρανού. Αλλά το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τις, με τις διαστάσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι άδικο. Και έχουμε και ένα πρόβλημα στην Ολλανδία, ιδιαίτερο. Πολλοί γεωργοί μας στις κάτω έχουν επενδύσει σε υποδομές, έχουν γύρει κτίρια, στάβλους και τώρα ισχύει μια γελία τιμή αναλυτρογάλακτος. Πώς θα αποσβέσουν τις επενδύσεις τους αυτοί οι άνθρωποι. Θυμάστε τι έγινε με τη Volkswagen και το σκάνδαλο. Τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά το θέμα είναι πόσο καιρό θα χρειαστεί η βιομηχανία για να διορθώσει την κατάσταση. Γιατί μπορεί να έχει χρόνο, αλλά νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι λάθος εδώ. Και για την κοινή πολιτική, Έχουμε ένα παράδειγμα με τη δική μου πατρίδα τη κάτω αλλά υπάρχουν και άλλε χώρε και εκεί θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερο διάστημα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα είναι πολύ πιο χρονοβόρα διαδικασία. Και επαναλαμβάνω, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι έχουν κάνει επενδύσεις, έχουν χτίσει κτίρια, αποθήκες ή σταθμούς για την επεξεργασία της κοπριάς. Θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο τώρα για να αποσβέσουν, να τι αυτές τις επενδύσεις. Ευχαριστώ κύριος Ντές. Yeah, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κόρτεν για την έκθεση, για την παρουσίαση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θέλω να αμφισβητήσω φυσικά τις καλές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το άρθρο 222 της συνθήκης που επεσήμαναν οι συνάδελφοι ε, δεν λειτουργεί με σύστημα εκούσιο. 50% στον ε, συνεταιρισμό, 50% στην ελεύθερη διάθεση έχουμε αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν πάει ο συνεταιρισμός για να πει «Α, πρέπει να μειώσετε κατά 50% την παραγωγή», ε, θα πρέπει να δώσετε και τη σχετική αποσημείωση. Και βεβαίω ο ιδιωτικό τομέα θα χαρεί ιδιαίτερο για αυτόν τον περιορισμό τη παραγωγή. Υπάρχουν γαλακτοκομικέ μονάδε οι οποίε έχουν στηριχθεί πάνω σε επενδύσει σοβαρέ και πρέπει να αποσβέσουν. Και αν οι άλλοι συνεχίσουν να παράγουν περαιτέρω, δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Με εκούσιο λοιπόν, με εκούσια δέσμευση, με αυτοδέσμευση δεν λειτουργεί το σύστημα. Πρέπει όλα τα κράτη, Γαλλία, Πολ, ε, Πολωνία, κατοχώρες ε, να μειώσουν όλοι την παραγωγή. Δεν μπορούν να μειώσουν δύο-τρία κράτη και οι άλλοι να συνεχίσουν να παράγουν όπως πριν. Το 222 λοιπόν από την οργάνωση αγοράς δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Και θα ήθελα όπως ανέφερε και η κυρία Μίλλερ να πω ότι θα είχαμε κύριε Κόρτε τη δυνατότητα με 200 εκατομμύρια ευρώ και με το, με τη μετατροπή του γάλακτο σε βούτυρο και ενδεχομένως ε, παγωτό να διαθέταμε τις ε, πλεονάσους ποσότητες και να αποφεύγαμε και την εισαγωγή ε, λοιπόν από την Ινδονησία. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, υπάρχει και η πρόβλεψη για τα 500 εκατομμύρια και επιπλέον το θέμα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ευθύνη θα αναλάβει. Υπάρχουν και οι εθνικές ευθύνε πολλοί είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι που μου λένε αν δεν ήμασταν υποχρεωμένοι στις καλές εποχές να πληρώνουμε τόσο υψηλού φόρους θα είχαμε ένα μικρό απόθεμα, ένα μαξιλάρι για να περνάγαμε πιο εύκολα μέσα από την κρίση. Γι' αυτό νομίζω τα κράτη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη ώστε να μην επιβάλλουν τόσο υψηλή φορολογία στους παραγωγού. Και ξέρουμε ότι δεν έχουμε αρμοδιότητες στον κοινωνικό τομέα, αλλά πρέπει πιστεύω κονδύλια του τομέα της γεωργίας να στραφούν και προς την κοινωνική υποστήριξη των γεωργικών οικογενειών. Έχουμε παραδείγματι ε, παραγωγούς στην ε, Γεωργία οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ψηλές ε, εισφορές να πληρώνουν. Ένας μισθωτός θα πληρώσει κατά το ίμιση τις δικές του εισφορές, το άλλο ίμιση θα το καλύψει ο εργοδότης του. Ο γεωργικός παραγωγός όμως πρέπει να καλύψει 100% τις εισφορές του. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να στηρίξουμε και με βέβαια με τα μέτρα και την παρέμβαση που αναφέραμε. Ο Επίτροπος Τσόλος είχε μιλήσει για 30.000 τόνους βούτυρου Ασήμαντη ποσότητα με 250.000 τόνους τώρα που γίνεται λόγος ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να ε, παραχθούν, αν και δεν βρήκε αυτό πλειοψηφία, νομίζω καταλήξαμε τελικά σε 70.000 τόνους, θα είχαμε ίσως τη δυνατότητα να απορροφήσουμε μεγαλύτερες ε, ποσότητες. Αγαπητέ Μάρτιν Χόισλινγκ, ξεκάθαρα δεν είναι δυνατόν να παρεμβαίνουμε χωρίς όριο, αλλά το να τραβήξουμε 150.000 τόνους ε, Ε, βούτυρο από την αγορά της Ευρώπης ε, θα σήμαινε αντίστοιχα και τη δυνατότητα να επιβληθεί η φορολογία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει καθόλου φορολογία, αλλά το βασικό είναι πριν ε, πέσουν πάρα πολλοί οι τιμές να γίνει αυτή η επέμβαση. Δεν μπορούμε να περιμένουν αυτά στα βάραθρα οι τιμές για να γίνει η επέμβαση. Αλλιώς, δεν πρόκειται να λειτουργήσει η αγορά. Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Κόρτε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παρουσίαση που μας έκανε. Εγώ, όπως και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι κατά τη γνώμη μου σωστό σε μια τέτοια κρίση την οποία θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, γιατί όντως ε, η Ευρωπαϊκή Γεωργία διανύει μια πολύ σοβαρή κρίση, αλλά θα πρέπει να ρίχνουμε το μπαλάκι στα κράτη-μέλη και να τα αναγκάζουμε να δώσουν μια λύση. Δεν θα πρέπει να μεταφέρετε τις ευθύνες στα κράτη-μέλη και να πληρώνουν ε, οι χώρες τα σπασμένα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε, να αναλάβει τα ενία της κατάστασης. Για το Γάλα, για παράδειγμα, τέτοιες αποφάσεις ε, και το άρθρο 222 θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά αν μια λύση είναι πανευρωπαϊκή, αν γίνεται και εφαρμόζεται παντού. Γιατί ξέρω ότι είναι οικειοθελής, προαιρετική λύση, αλλά αν δεν γίνεται ταυτόχρονα το μέτρο από όλου, τότε δεν θα έχει νόημα. Εγώ κατάγομαι από την Ισπανία, από μια χώρα που παράγει πολύ λιγότερο γάλα από ό,τι καταναλώνει. Και ήδη έγινε πριν από δεκαετίες μια ε, αλλαγή στον τομέα και στροφή σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς. Παράγουμε λοιπόν πολύ λίγο γάλα, λιγότερο από ό,τι καταναλώνουμε, αγοράζουμε δηλαδή γάλα από άλλε χώρε μέλη και τώρα η Ισπανική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που είναι γενικό ε, προτείνοντας μία μείωση σε μία πενταετία της παραγωγής του γάλακτος γύρω στο 2%. Ενώ ήδη η παραγωγή μας είναι χαμηλή και ήδη κάναμε μία μεταστροφή προς άλλους τομείς. Δεν είναι καλό ο προσανατολισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή σε μία τέτοια που είναι γενική, που είναι ε, πανευρωπαϊκή και είναι κρίση ευρωπαϊκής γεωργίας, η λύση που εμείς διαλέγουμε να είναι η λύση που υιοθετούμε σε πολλές άλλες αποφάσεις, η λύση της επανεθνικοποίησης. Δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο και αφιβάλλω είναι και αποτελεσματικό γιατί δυστυχώς κατά πάσα πιθανότητα ούτε και αυτό το μέτρο που προτείνεται θα, φέρει, θα αποφέρει καρπούς. Μερικές χώρες ε, μπορεί να είναι διατεθειμένες, ε, αλλά είμαι πολύ επιφυλακτική, έχω φοβερούς ενδιασμούς για το μέτρο. Το μέτρο είναι καλό, αλλά θα είναι αποτελεσματικό μόνο αν υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη, ταυτόχρονα και ισχύσει για όλους. Κύριε Κόρτα, έχω και μία ερώτηση. Αναφερθήκατε στην παράταση των ε, ενισχύσεων ε, για το ρωσικό εμπάργο. Από ό,τι είπατε, ε, είναι διαθέσιμα λιγότερα κονδύλια, λιγότεροι πόροι. Οπότε ρωτώ, θα εξασφαλιστεί μια συνέχεια ή μήπω θα υπάρξει διακοπή για ένα διάστημα των ενισχύσεων. Γιατί η παράταση θα έχει νόημα να είναι άμεση, να μην δημιουργηθεί κενό ή χάσμα και να μην επηρεαστούν ε, παραγωγές απορροκυπευτικών. Να μην υπάρξουν κενά στην παράταση. Και τελευταία ερώτηση. Γιατί τα κράτη-μέλη ε, δεν δαπανούν σε μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης αυτά τα 500 εκατομμύρια που προβλεπόταν στο πακέτο αντιμετώπιση τη κρίση του Σεπτεμβρίου. Πού είναι το πρόβλημα, γιατί τα κράτη-μέλη δεν εκταμιεύουν τα χρήματα αυτά. Τι συνέβη. Ευχαριστώ. Κύριο Σφερό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα έλεγα από τι συζητήσει μα αυτό που προκύπτει είναι πολύ κακό για το τίποτα. Το Μάρτιο του 2015 όλοι δεχτήκατε εδώ την απορρίθμιση του τομέα του γάλακτο και το τέλο των γαλακτοπαραγωγικών ποσοστώσεων. Τέλο πάντων, οι περισσότεροι έστω. Οι περισσότεροι, διότι οι περισσότεροι εκτό από κάποιου ε, από του αντάρτε του γαλατικού χωριού ήσασταν σύμφωνοι. Και μετά έρχεστε ένα χρόνο μετά να μα πείτε θα περάσουμε σε διαπιστώσει. Ποια είναι η διαπίστωση. Ένα χρόνο μετά την απορρίθμιση, το Μάρτιο του 2015 δηλαδή, είμαστε σε κρίση. Την κρίση αυτή μπορούσαμε να την έχουμε προλάβει. Να την έχουμε προβλέψει. Μία είναι η βούληση που έχουμε ε, πλέον Μάλλον, αυτό που θέλατε να περάσετε ήταν ε, να πιέσετε σε μία αλλαγή και να καταστρέψετε ένα τομέα, ενώ τώρα αυτό που θέλουμε να επιστρέψουμε την εθνική κυριαρχία και κάθε χώρα να επανέλθει στο παλιό καθεστώ για τον τομέα του γάλακτο. Μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα υπάρχει κρίση, ότι η επιτροπή Χόγκαν ε, τα γρυπνεί. ώστε να υπάρχει μια αξιοπρεπή γαλακτοκομική παραγωγή στην Ευρώπη. Εγώ έχω να θέσω ένα ερώτημα εδώ στην Ευρωπαϊκή Παραγωγή. Μας έχει υποβληθεί ένα πρόγραμμα που δεν είναι πρόγραμμα για τις χώρες που θέλουν να αυξήσουν την γαλακτοκομική τους παραγωγή. Μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή αυτή ε, κάνοντας και αποθήκευση, διότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, το έκτακτο πρόγραμμα μέτρων ε, της Επιτροπής ε, του κ. Χόγκαν χάνει κάθε θεμητό και κάθε σκοπιμότητα. Διότι κάποιοι με αυτή την άποψη της παραγωγής θα θεωρήσουν ότι κάποιοι θα πάψουν ε, να παράγουν μόνο και μόνο για να καταλάβουν μερίδια στην αγορά. Αυτό είναι ουσιαστικά μια παροδία. Ο μόνος σας στόχος είναι με τρόπο ηθελημένο και οριστικό να οδήγησετε την Ευρώπη προς τον άκρα του φιλελευθερισμό. Αυτό είναι όλο. Ευχαριστούμε κύριο Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Κύριε Κόρτε, αλλά είπατε τρεις λόγους για τους οποίους μπορεί να έχουμε κρίση μιλήσατε για την καταπίεση των, ε, τομέ, των, των τιμών, την πτώση των τιμών διεθνώς και το ρωσικό εμπάργκο. Ένα τομέα που δεν αναφέρατε είναι εξή. Είναι πολύ εκτός του γεωργικού κλάδου αυτοί που δεν λερώνουν ποτέ τα χεράκια τους και δεν θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν μια γελάδα από ένα άλλο ζώο που θέλουν να βγάλουν λεφτά, ε, να λαιλατίσουν τον τομέα αυτό και ενώ συνεχίζουν να το κάνουν ε, και θέλω να φάνε διαμιά σε όλη την τούρτα αντί να την κόβουν σε φέτε. Και αυτό νομίζω το καθένα μπορεί να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται να ή σεφ. Ε, δεν λειτουργεί. Καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα. Ε, φαίνεται ότι κάποιοι είναι απελπισμένα άπλιστοι. νομίζω λοιπόν ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αρμέγουμε τι ίδιε αγελάδε. Δείτε τι γίνεται στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή, όπου οι εκτροφεί δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν. Όμως, αυτό που αρχικά θα τους βοηθούσε, οι συνεταιριστικέ κινήσεις ε, και οργανώσεις έχουν καταλήξει σε τέρατα. Τέρατα όπου ενώ υπάρχει κρίση η ΚΟΑ λόγου χάρη που θα βοηθούσε τους γεωργούς και την κοινότητα τα τελευταία δύο χρόνια αποφάσισε να πληρώσει τα εννέα εκτελεστικά της ελέγχη 9.000 ευρώ μισθό στον καθένα. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. 5.000 ευρώ χάνονται καθημερινά τα τελευταία δύο χρόνια για κάθε κτηνοτρόφο και γαλακτοπαραγωγό στην Ιρλανδία. Το ίδιο και στον τομέα του Βόλου. Δεν φαίνεται να μπορούμε να αποκομίσουμε κερδό, αλλά εδώ ένα Ιρλανδό ανακοίνωσε κέρδη 52,6 εκατομμύρια ευρώ σε μια από τις εταιρείες του που έχει σύνδεση με την ABP. Αυτοί δεν λερώνουν τα χέρια τους, ούτε αγγίζουν τις αγελάδες προφανώς, αλλά έχουν καταφέρει να έχουν τεράστια κέρδη. Και επιπλέον δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν παρά μόνο τα ανώτατα στελέχη και τους φόρους. Ακούτε, 152.000 ε, και 52 εκατομμύρια. Πραγματικά, με όλες τα σχέδια και τα προγράμματα, Πώς περιμένετε να πάρουν όλοι ένα κομμάτι από το γλυκό, ε, αν υπάρχει ένας τεράστιος χοντρός στην άκρη του τραπεζιού, ο οποίος κάθεται και τρώει όλο το γλυκό μόνος του. Πώς θα συνεχιστούν αυτά, αν συνεχίσετε κατά αυτόν τον τρόπο, αν βιτρίσετε ε, αυτή τη στάση. Οι γεωργοί δεν παίρνουν τίποτα στα χέρια τους και αυτό δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, διότι οι άνθρωποι εκτός του γεωργικού κλάδου κερδίζουν εκατομμύρια και αυτοί που κάθονται και υδρώνουν και δουλεύουν, χάνουν λεφτά και ουσιαστικά αυτοκτονούν. αυτοκτονούν. Τι σα εκπλήσει όλο αυτό. Ο κύριος Δεκάστρο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Υπόθηκαν ε, πολλά. και άκουσα και τι τελικές σας σα Κύριε Κόρτα, σα ευχαριστούμε. Στην ανάλυση σας δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα, αλλά το πρόβλημα είναι πώ να διαχειριστούμε την κρίση αυτή. του άρθρου 152 είναι ένα εργαλείο που εθελοντικά δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Προκαλεί σοβαρότατε στρεβλώσει και το θύμισε και η συνάδελφο Αγγιλέρα στην Ισπανία λόγω χάρη και στη δική μου χώρα. Ανάλογη κατάσταση. 40% του γάλακτο το εισάγουμε. Η παραγωγή ελέγχεται πλήρω από το κεντρικό επίπεδο. Πώ θα συνεχιστεί αυτό. Ε, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αλλά μόνο μια ευρωπαϊκή λύση μπορούμε να έχουμε και πρέπει να βρούμε τρόπους να ελέγξουμε την προσφορά. Ο κύριος Νταντά το είχε πει και στη, στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ε, επέστρεψαν παλιά επιχειρήματα, όντως κύριε Νταντά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε τη σωστή αλλαγή. 500 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική οικονομική συνεισφορά, αλλά τελικά διανεμήθηκε στα κάτι μέλη χωρί να υπάρξει καμία αποτελεσματικότητα ή έστω χωρί να χρησιμοποιηθούν σωστά. Ε, Προ στιγμή, οι επιλογέ τη Ευρώπη για να επιληθεί το πρόβλημα ε, υπερισχύουν των εθνικών. Ευχαριστούμε κύριο Γιάρ. Ναι, Πρόεδρε, θα ήθελα να διορθώσω μερικά πράγματα. Καταρχάς, το μέγεθος επιχείρησή μου, 400 εκτάρια μαζί με άλλου που συνεργαζόμαστε. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να είχαμε και 2.000 εκτάρια, αλλά δεν τα καταφέρνουμε όλα. Και επίσης δεν έχω ούτε γάλα, ούτε γουρούνια και άρα άμεση συνάφεια με τα θέματα που συζητούμε και συμφέρον δεν έχω. Όταν ε, λοιπόν είναι αναγκαία μια κοινωνική πολιτική σε εποχές δύσκολες, σε εποχές κρίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχόμαστε ότι είναι αναγκαία μια ευρωπαϊκή πολιτική και σε καλές θα χρειαστούν λοιπόν περισσότερα κονδύλια για την στήριξη του κάλακτος. Για το 2017 φαντάζομαι ότι ενδέχεται να μην υπάρχει καμία δυνατότητα αύξηση των δαπανών. Ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια διόρθωση βέβαια στον προπολογισμό. Θα πρέπει ξεκάθαρα να επισημανθεί ότι υπάρχει ανάγκη για μια πιο ευέλικτη διαχείριση κρίσεων, γιατί το σύστημα δεν μας επιτρέπει να ε, δώσουμε λύσεις και ίσω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε στον προπολογισμό γιατί αν υπάρχουν προβλήματα δεν είμαστε θέση να δώσουμε οποιαδήποτε υποστήριξη στον γεωργό ή στον κτηνοτρόφο. Επίσης, ε, το επισήμανε πολύ καλά η στον τροφο Επίση, το επισημανε Μιούλερ, το γαλακτοκομείο δεν είναι απαραίτητα ο εταίρος με τον οποίο θα συνεργαστούμε, γιατί μπορεί να θέλει να συνεργαστεί, μπορεί να μην θέλει να συνεργαστεί βεβαίως πιστεύω ότι θα πρέπει κάθε λίτρο γάλακτος να πληρώνεται στην ίδια τιμή ανεξαρτήτως της, ε, του προορισμού στον οποίο κινείται. Το ίδιο ισχύει με τα σιτηρά. Ορίζω μία τιμή και ανεξαρτήτως της ποσότητας αυτή η τιμή πάει η ίδια σε όλους. Το ίδιο πρέπει να ισχύει λοιπόν και το γάλα για κάθε παραγωγό να ισχύει η ίδια Βεβαίως ένα ζήτημα θα μπορούσε να είναι το ζήτημα της φορολογίας ή κάποιες ε, πληρωμές για τιμές στόχου. Χαίρομαι που δεν έγινε λόγος για ποσοστώσεις. Ας είμαστε και λίγο σοβαροί. Έχουμε αντιμετωπίσει εξαιτία των ποσοστώσεων στο γάλα αρκετές κρίσεις στο γαλακτοκομικό τομέα. Θεωρούσαμε ότι θα ήταν ε, ε, το Ζαναντού αυτή η λύση των ε, ποσοστώσεων στο γάλα. Θα μας έδινε λύση σε κάθε μας πρόβλημα, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις. Και νομίζω Καταλαβαίνοντα βεβαίω ότι η Ευρωπαϊκή Επίτροπη δεν θέλει να λάβει μέτρα για περιορισμό των ποσοτήτων, γιατί ταυτόχρονα πιστεύει ότι η οργία, οι κτηνοτρόφοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν τι σχετικέ πρωτοβουλίε και άρα δεν θέλει να προχωρήσει του περιορισμού και καλεί τα κράτη-μέλη να αναλάβουν, να εμπλακούν στην υπόθεση αυτή. Αλλά νομίζω τότε γίνεται ακόμα πιο χαοτική η κατάσταση και γι' αυτό απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντα να προτείνει ευρωπαϊκές λύσεις, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για το πώς μπορούν να περιοριστούν οι ποσότητες, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει, να δοθεί κάποια λύση. Ίσως η αξιοποίηση, ίσως η ε, διάθεση σε άλλους τομείς για μεταπίεση να ήταν μια λύση. Δεν μπορούμε να μετακυλούμε το πρόβλημα με την αποθήκευση μόνο των ποσοτήτων, των ποσοτήτων. Βεβαίως ένα ζήτημα είναι το εμπάργκο της Ρωσίας, πρέπει να βρούμε λύσεις γι' αυτό. Και ίσως πρέπει να κοιτάξουμε και τους λόγους πίσω από αυτό το εμπάργκο. Για όσους ζητούν την κατάργηση του Υπουργό Γεωργίας της Ρωσίας βρίσκεται σε, ένα μαύρο, μια μαύρη λίστα. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα και κατά τα άλλα πρέπει να δώσουμε λύσεις που να ισχύουν για όλους. Ευχαριστώ κύριε Σεβαστιά. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για ένα τομέα, το τομέα των όποροκυπευτικών, ε, για, το, τον οποίο η κρίση είναι χρόνια, όχι προσωρινή. Και μάλιστα οι προοπτικές είναι πολύ ζωφερές. Και δεν το λέω αυτό εγώ, αλλά η έκθεση μέλο που εγκρίναμε και στην Επιτροπή μας, αλλά και στην Ολομέλεια. Και οι, οι λόγοι είναι σαφείς, τα αίτια είναι σαφή. Α, αθέμετους ανταγωνισμούς από τρίτε χώρε χωρί να πληρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής, ούτε οι περιβαλλοντικές, ούτε οι υγειονομικέ, ούτε οι εργασιακέ και ταυτόχρονα έχουμε τι πιέσει από τι μεγάλε αλυσίδες διανομή. Όλα αυτά είναι γραπτά, τα γνωρίζουμε, τα συζητήσαμε άπειρε φορέ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τολμά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και οι συνέπειε είναι γνωστέ. Εγκατάλειψη των γεών, χιλιάδε εκτάρια εγκατάλειψη κάθε χρόνο, κυρίω στην Νότια Ευρώπη και η γύρανση του γεωργικού πληθυσμού. Σε 15-20 χρόνια δεν θα έχουμε πια ε, παραγωγούς οποροκυπευτικών στην Νότια Ευρώπη. Βέβαια, αν ε, πεθάνει το σκυλί, πάει και η λύσα. Έτσι θα χαθεί και το πρόβλημα. Είναι μια παροιμία που έχουμε στην Ισπανία. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Επίση, έχουμε το ρωσικό εμπάργκο. Με προβληματίζουν οι διασμοί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την παράταση μέσω κατεξοδότηση πράξη των έκτακτων μέτρων. Ο κλάδος ζητά όχι μόνο παράταση των μέτρων αυτών, αλλά και πιο αποτελεσματικά μέτρα. Για παράδειγμα, μια και έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερωτώ, θα επισέλθουν και άλλα προϊόντα στο θέμα, όπως η λωτή ή τα ρόδια που δεν καλύπτονταν αρχικά από τα μέτρα και παρόλα αυτά είχαμε και στα προϊόντα αυτά ρόδια και λωτούς ε, κατάρρευση των τιμών. Ερωτώ λοιπόν, θα θεσπιστεί επιτέλους η παράταση και αν ναι πότε και θα είναι άμεση εφαρμογή. Γιατί για τα, για τα γλυκά καλοκαιρινά φρούτα η παραγωγή ε, είναι πολύ ανήσυχοι, τους έχουν ζώσει τα φίδια για το τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση ή δεν συμπεριληφθούν και νέα ε, προϊόντα. Επίσης, ε, ισχύουν οι μηχανισμοί πληρωμής για τα προϊόντα που δεν υπόκειται στην απόσυρση και δεν χρησιμοποιούνται ε, τα μέτρα αυτά γιατί οι τιμές είναι τόσο εξευτελιστικές που δεν συμφέρει ούτε η συλλογή ε, των καρπών ε, για τους γεωργιούς και μάλιστα δεν τους συμφέρει να προσλάβουν και κόσμο για να κάνει τις δουλειές αυτές γιατί ούτε καν ε, την συλλογή δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν για να μην μιλήσουμε για μεταφορά. Τώρα, οι μεταποίησεις που γίνονται και η επεξεργασία προκειμένου να γίνουν ε, πουρέδες, ε, χυμή κτλ. Ούτε και αυτά αξίζουν, συμφέρουν. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να καταβληθεί μια αξιοπρεπή τιμή για τα προϊόντα αυτά. Γιατί το καταλαβαίνουμε ότι ήταν ε, σημαντικό να πληρώσουμε με κυρώσεις στη Ρωσία, η οποία υιοθέτησε ως αντίπεινα το εμπάργο, αλλά τελικά τα σπασμένα από όλη την κατάσταση αυτή την πληρώνουν οι γεωργοί που ήδη έχουν τιμωρηθεί αρκετά νομίζω. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και συζητούμε για το θέμα αυτό, ας μην ξεχνούμε ότι ο βασικός λόγος ε, της κατάρρευσης των τιμών ε, ε, πέραν της, του ρωσικού εμπάργου των αθέμητων, των ανταγωνισμών από την Κίνα, ξεχάσαμε και τη μείωση των τιμών πετρελαίου και ταυτόχρονα εκατομμύρια ανθρώπους, εκατοντάδες εκατομμύρια που ακριβώς επειδή τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί δεν έχουν αρκετά για να αγοράσουν το τρόφιμα και να επενδύσουν στη διατροφή τους. Όλα αυτά οδήγησε και σε μείωση της κατανάλωσης. Και δεν φταίνε για όλα αυτά οι γεωργοί. Δεν είναι οι γεωργοί οι πέτοι της κρίσης. Ήταν κυρίως πολιτική και οικονομική οι λόγοι της κρίσης αυτής, την οποία πληρώνουν όμως οι γεωργοί. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν μια ε, κατάρρευση των τιμών και τώρα καλούμαστε να συζητήσουμε για τις ενισχύσεις προς τους γεωργούς. Και εγώ σε αγροτική εκμετάλλευση μεγάλωσα, σε έναν οπορώνα με παραγωγή μήλων και μπορώ να πω ότι από το προσωπικό μου βιώματα ότι οι γεωργοί δεν θέλουν ε, ελεημοσύνη, δεν θέλουν βοήθεια. Θέλουν να μπορούν να επιβιώνουν, να βγάζουν τα ζήν με τον υδρότο του προσώπου τους. Και δίνεται η εντύπωση ότι οι γεωργοί ζητούν την ενίσχυση και επιπλέον κατηγορούνται για την περιβαλλοντική ρήπαση. Ενώ όλοι γνωρίζουμε πόσο ζωτικό είναι ο ρόλο τη γεωργία. Είναι πολύ άδικη η κατάσταση αυτή για του γεωργού. Και πολύ συχνά οι γεωργοί είναι και τα θύματα πολιτικών παιχνίων. Βλέπε ρωσικό εμπάργο. Και μπορώ να σα πω από την προσωπική μου πείρα τι συμβαίνει στη Σλοβενία. Εκεί η βασική γαλακτοπαραγωγική εταιρεία αγοράστηκε από τη γαλλική εταιρεία Λακτάλης και σε αρχές Απριλίου η εταιρεία αυτή έλαβε συμβάσεις από τον αντίστοιχο συνεταιρισμό ζητώντας μείωση της παραγωγής γάλακτος, ήδη δηλαδή με, με το τερματισμό των ποσοστώσεων και επίση ανέλαβε τη δέσμευση ότι αν δεν μειώσει την παραγωγή θα υποστεί κυρώσει 50 λεπτά το λίτρο. Φανταστείτε, με ήδη χαμηλέ τιμέ, μια επιπλέον ποινή, ένα επιπλέον πρόστιμο, τι πλήγμα είναι για το συνεταιρισμό αυτό εν μέσω κρίσης και με τόσο χαμηλές τιμές. Και οι χώρες που έχουν τις αλυσίδες παραγωγής, αλυσίδες επεξεργασίας και τις μεγάλες αλυσίδες διανομής που λύνουν και δένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε καλύτερη μοίρα. Αλλά οι πιο νέες χώρες που η γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι καλά οργανωμένοι, υφίστανται ακόμη πιο έντονα τις συνέπειες της κρίσης. Και αναγκαζόμαστε να αγοράσουμε γεωργικά προϊόντα από άλλες χώρες που έχουν πιο ανεπτυγμένη γεωργία. Και αυτό, αυτό που μου προέχει είναι να μειώσουμε την παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι ο καθένας όπου θέλει. Αλλιώς δεν πρόκειται να επιλύσουμε το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ενισχύσεις ε, προς τους γεωργούς. Ξέρω το σλοβενικό πρόγραμμα ε, που ήταν επιφορτισμένο με την κατανομή των ενισχύσεων προς γεωργούς. 37 ευρώ αναγελάδα το χρόνο ήταν στη Σλοβενία το πρόβλημα και με παρούσα τιμή 36 λεπτά ε, το λίτρο σημαίνει ότι η ενίσχυση θα κάλυπτε 150 λίτρα γάλακτος ουσιαστικά. Ενώ οι παγκόσμιες τιμές έχουν, ε, του γάλακτος έχουν μειωθεί κατά 35% που σημαίνει ότι ε, οι κτηνοτρόφοι, οι γαλακτοπαραγωγοί έχουν υποστεί τεράστιε ε, ζημιέ εξαιτία τη μείωση τη τιμή γάλακτος. Μπορούμε να θεσπίζουμε ενισχύσει, αλλά δεν πρόκειται να αποζημιώσουμε ποτέ του γαλακτοπαραγωγού για τι τεράστιε ζημιέ που υπέστησαν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή τιμή γάλακτο για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι γαλακτοπαραγωγοί και να συνεχίσουμε να έχουμε γαλακτοκομικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά είναι αργή στην αντίδρασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα φλεγής, Εγώ παρακολούθησα τις συζητήσεις από την αρχή και συμφωνώ με κάποιους συναδέλφους που είπαν ότι μόνο καθυστερημένα ξύπνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνειδητοποίησε την κρίση που διανύουμε όταν οι, οι διαστάσεις ήδη έγιναν ανεξέλεγκτες. Χρειαζόμαστε κατάλληλου μηχανισμού που να μας επιτρέπουν πανευρωπαϊκά να μειώσουμε την παραγωγή και ταυτόχρονα να θεσπίσουμε μια αποζημίωση για να εγγυηθούμε φυσιολογικέ τιμέ προς τους ε, αγρότε μας. Αυτό θέλουν, φυσιολογικέ τιμέ και προτιμούν τέτοιες τιμέ παρά να περιμένουν την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στα απορροκυπευτικά παρόμοιες εξελίξεις διαπιστώσαμε. Είχαμε μία διετία αποσύρσεων από την αγορά, χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων φρούτων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και μάλιστα επειδή το εμπάρκο που ξεκίνησε τον Αύγουστο καθυστέρησε κάπως ο αντίκτυπος. Αλλά είχαμε πρόβλημα μετά στη Σλοβενία και την Πολωνία και η μεγάλη παραγωγή μείωσε ακόμη περισσότερο τις τιμές με αποτέλεσμα οι γεωργοί να λαμβάνουν πολύ χαμηλά ποσά εξαιτία του κορεσμού που επικράτησε στην αγορά των απορροκευτικών. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση, να έχουμε επίγνωση των διαστάσεων της κρίσης και να θεσπίσουμε κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Οι ΔΕΜΗ θα κατεβάσουν τα ρολά οι γεωργοί σε, λίγο, σε λίγους χρόνους και θα χάσουμε το γεωργικό μας τομέα. Θα πρέπει να επανεφεύρουμε το μοντέλο μας και να επενεκκινήσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένας δρόμος με επιστροφή. Αν κλείσει μια γεωργική επιχείρηση, πολύ δύσκολα θα ξανανοίξει. Ευχαριστώ κύριο Άγγινιου. Πρόεδρε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα τόσο πολύ στη συνεδρίαση, ήταν αναπόφευκτο. Μιλάμε για τι κρίσει στη Γεωργία, όμω οι περισσότεροι και οι προλύσαντες Κυρίω μίλησαν για το γαλακτοπαραγωγικό τομέα. Αυτό όμω ο τομέα φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ δύο στενών. Πρώτα απ' όλα, από τη μια έχουμε μια τελείως εθνικοποιημένη γαλακτοπαραγωγική βιομηχανία και εδώ νομίζω ότι μιλάτε για ένα εξευρωπαϊσμένο γαλακτοπαραγωγικό τομέα. Ε, λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χειρίζεται όλα από την εθνική από την άλλη, θα πρέπει να διαλέξουμε αν θέλουμε μία βιομηχανία που να την οδηγεί η ίδια η παραγωγή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ των δύο. Και ότι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει η πολιτική είναι ότι την αγορά θα τη διαμορφώσει η ίδια η βιομηχανία. Δεν υπάρχει ένα κλασικό γαλακτοπραγωγό. Μπορεί να είναι κανεί γαλακτοπραγωγό έχοντα 10 γελάδε, αλλά μπορεί να έχει και 30. προστιθέμενη αξία μπορεί να έχει κάθε σταγόνα γάλακτο που παράγει. Κάποιοι, όπω στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κτηνοτρόφοι, έχουν πάνω από χιλιάδε γελάδε. Μιλάμε για τεράστιε επιχειρήσει, δεν μιλάμε για του γελαδάριδε με ε, το σανό και την, ε, για το γκουβά, για το γάλα. Εδώ λοιπόν, εάν δούμε έναν άλλο τομέα, αυτόν που έχει απασχολήσει ιδιαίτερο σε μένα λόγω χάρη, την παραγωγή των αυγών, δεν έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ακόμη η πολιτική με την καθορισμό των τιμών. Ο ίδιος ο τομέας μπορεί να ε, διαχειριστεί τα προβλήματά του. Πριν από 30 χρόνια περίπου υπήρχαν ε, παράπονα ότι η βιομηχανία είναι όλο και πιο αποτελεσματική. Οι καταναλωτές είχαν ε, πρόβλημα με την παραγωγή αυγών, αλλά οι παραγωγοί κυρίσαν και του εξήγησαν ότι αν θέλετε φθηνά αυγά, αυτό είναι ο τρόπος να τα παράγουμε. Αυτή είναι η μέθοδος παραγωγής. Αυτόν τον τομέα λοιπόν τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η ίδια η βιομηχανία βιομηχανία, οι ίδιε οι επιχειρήσει. Μόνοι του έχουν ορίσει τα πρότυπά του, μόνοι του έχουν ορίσει τι υποθεωρήσει του και του ελέγχου του. Και εδώ βλέπω τα πρώτα φώτα, τι πρώτε αναλαμπέ ενό απελευθερωμένου τομέα γάλακτο. σω αυτό να ήταν μια λύση, αλλά να προσέξουμε, διότι τα σούπερ μάρκετ μα λένε ότι οι καταναλωτέ δεν θέλουν να διαρκώ διοικημένε τομέ τιμές, απ' την άλλη η παραγωγή μας λένε ότι θέλουν να παράγουν με τιμή επικερδή, αυτό που βλέπουμε ε, είναι είτε έναν απελευθερωμένο τομέα γάλακτος, είτε έστω ε, ελεγχόμενες τιμές. Δηλαδή κανείς ε, προσυπογράφει σε ένα συνολικό πρόγραμμα και τα σούπερ καταβάλουν μια φίξ τιμή. Αυτός είναι ένας τρόπος. Θα μπορούσε κανείς να ακολουθήσει και άλλο εδώ. Θα ήθελα πάντως να δω τα κάτι μελη και ιδίως το δικό μου όταν πρόκειται για αυτά τα μικρά κοπάδια λόγου χάρη να λένε ωραία θα σας δίνουμε ένα συγκεκριμένο ποσό για να ε, προσεχθείτε εξωπρεπώ. Πάρτε αυτό το ποσό, μην ξαναπαράγετε σταγόνα γάλακτο, αλλά αν θέλετε ένα άλλο πρόγραμμα ή την προστασία του περιβάλλοντο ή κάτι άλλο, κάτω τι θέλετε, απλώ μην παράγετε γάλα. Μην παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να επιβιώσετε. Αυτέ είναι ορισμένε ιδέε που ήθελα να σα ρίξω έτσι στο τραπέζι τα αποστοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή τι ακούμε, γκρίνια, γκρίνια και γκρίνια και τελικά δεν είναι αυτό η λύση. Merci, Madame Maguinness. Ευχαριστούμε. Να συμφωνήσω κι εγώ, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να με καθυστερήσουμε, δεν εξαρτάται από εμά. Ε, τώρα να συνεχίσω από εκεί που ε, άφησα το θέμα ο ε, για την διεθνή προσφορά. Με ενδιαφέρει πολύ και αυτό με ρωτάνε οι κτηνοτρόφοι μας, όχι ακριβώς τι ισχύει το, για το άρθρο 22, αλλά ποια είναι ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα στοιχεία που έχετε, τι προβλέπετε για την αύξηση παραγωγής της ΗΠΑ λόγω χάρη και πότε η τάση αυτή ενδεχομένως θα αλλάξει. Είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ε, συνεχίζοντας από αυτό, οι μέρημνες που ακούστηκαν και από άλλους, η υλοποίηση του άρθρου 222. Πώς θα ε, λειτουργήσει στην πράξη αυτό. Ίσως πρέπει να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα, να το δούμε στην Επιτροπή αυτή, στην Ολομέλεια, ποια είναι η διαδικασία που να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Έχει γίνει αποτίμηση, εξολόγηση μάλλον της ε, πρόσληψης της πρότασης αυτής και οι τιμέ στην αγορά πώ θα επηρεαστούν ε, λόγω τη πρόταση. Και αυτό θα ήταν σημαντικό να το ξέρουμε. Διότι σε κάθε περίπτωση Υπάρχουν τεράστιε ανησυχίες για την κατάσταση στην αγορά, όχι μόνο για το γάλα, αλλά και για άλλε περιπτώσει ε, γεωργική παραγωγή. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε ποιε είναι οι μακροχρόνιε ε, προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Νταντά. Κύριε Πρόεδρε, πολλά υπόθηκαν ήδη. Και βλέπω ότι επιδεικνύει περισσότερη συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τοποθέτησή τη σήμερα παρά αυτό που είχε δείξει πριν από λίγου μήνε. Εγώ δύο ερωτήσει επιπλέον θέλω να θέσω στον κύριο Κόρτα. Πρώτον, να σκεφτούμε, νομίζω, την ε, χρήση, τη συνετή χρήση των χρημάτων μας. Δηλαδή, μπορούμε να βλέψουμε ένα σύστημα που να επιτρέπει ταυτόχρονα και στους ε, κτηνοτρόφους να καθορίζουν τις τιμές της αγοράς, αλλά και να καλύπτονται, να προστατεύονται οι πλέον ε, ε, ευάλωτοι, ευπαθείς. Κυρίως με την αύξηση των προσφύγων. λόγω χάρη, αν καταναλώνουν ένα λίτρο καθημερινά ανά άτομο, θα διπλασιάσουμε την παραγωγή μα. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι με την νομική μα βάση. Να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο έκτακτο. Σε έκτακτες συνθήκες απαιτείται και έκτακτο νομοθετικό πλαίσιο. Ή τα μέτρα πρόβλεψης μείωσης με σφαγή ε, γελάδων. Θανάτωση γελάδων. Εδώ προκύπτει ένα τεράστιο ζήτημα. Πριν από τρία χρόνια προβλέπαμε ότι η διεθνή ζήτηση θα αυξάνεται. Εάν αρχίσουμε να σκοτώνουμε τις αγελάδες θα χρειαστούν τέσσερα χρόνια, τρία, για να ξαναφτάσουμε στην σωστή γαλακτοπραγωγή. Ε, τέσσερα χρόνια είναι η οικειοφορία. Όταν ε, αρχίσουμε να σκοτώνουμε και Όταν αρχίζουμε λοιπόν να σκοτώνουμε τις ε, αναπαραγωγικές αγελάδες, πιθανώς να έχουμε και άλλα προβλήματα και με την παραγωγή του κρέατος. Αυτό να σκεφτούμε λοιπόν γιατί θα χρειαστεί μια τετραετία για να καλύψουμε αυτό το κενό. Ευχαριστώ. Έδωσα σε όλους το λόγο εκτενώς. Ε, θα προσπαθήσω ο κύριος Κόρτε να απαντήσει. Βλέπετε κύριε Κόρτε πόσοι συνάδελφοι παρενέβησαν. Βλέπετε τις εκκλήσεις που σας απευθύνθησαν και είναι σχεδόν ομόφωνες. Νομίζω είναι σημαντικό να συμφωνήσετε κι εσείς και ο Επιτροπός σας ότι αυτά πρέπει να λεφθούν σοβαρός υπόψη. Ε, χρειαζόμαστε τουλάχιστον κάποιες πρώτες ε, απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις πολυάριθμες ερωτήσεις που ετυπώθηκαν. Ίσως ενώνοντας τα σε διάφορα θεματικές ενότητες, ένα από τα πρώτα ζητήματα που ετέθησαν επίκριση σχετικά με το άρθρο 222, ότι δεν έφερε αποτελέσματα σε καμία περίπτωση και τι θα κάνει η Επιτροπή. Κοιτάξτε, η απάντησή μου Μπορεί να είναι γραφειοκρατική εκ πρώτη όψου, αλλά δουλεύουμε σε ένα σύστημα οργάνωση, κοινή οργάνωση αγορά. Αυτό είναι ο βασικό κανονισμό, βασική πράξη. Προβλέπει μια σειρά από μέτρα. Και άλλα μέτρα δεν τα, προσφέρει, δεν τα προβλέπει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αν μου πείτε, μπορεί να κάνει η Επιτροπή πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού, γιατί το σύστημα δεν λειτουργεί κτλ. Αλλά ακόμα αυτό δεν έχει κρυθεί νομίζω. Με το 222 για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε τέτοιο μέτρο. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε τέτοιο μέτρο. Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο που έδινε το γράμμα του κανονισμού και τώρα νομίζω ότι αντί να ε, βάζουμε την ετοιμιγωρία ότι δεν φέρνει αποτέλεσμα, θα ήταν καλό όλοι μας, Κομισιόν, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρει αποτέλεσμα και να απευθύνουμε αυτή την έκκληση και στον κλάδο και στα γαλακτοκομεία και τους συνεταιρισμού για τους οποίους τόσες επικρίσει ακούστηκαν να αξιοποιήσουν το σύστημα. Γιατί σε ένα σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν ποσοστώσει, θα πρέπει ο κάθε ε, ένας ή κάθε μία επιχείρηση εκμετάλλευση να λαμβάνει πλέον τι ευθύνε των αποφάσεών τη. Δεν έχει πλέον την εξουσία Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό ποσοστώσεων ή για ε, διατάγματα τα οποία θα απαγορεύουν την παραγωγή, ούτε και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν βεβαίω ένα τεράστιο περιθώριο πυθού. και μπορούν να καταστήσουν κατανοητό για τους πάντες ότι η κατάσταση που οδηγεί σε όλα αυτά τα προβλήματα στο γαλακτοκομικό τομέα είναι ότι παράγονται υπερβολικά μεγάλες ποσότητες γάλακτος σε ορισμένες περιοχές. Βλέπουμε μέχρι και 20% αύξηση στην παραγωγή τον τελευταίο χρόνο. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν. Χρήματα. Θα υπάρξουν άρα και χρήματα για να ενισχυθεί αυτή η δύναμη της πυθούς. Ο Επιτροπός είπε στο Συμβούλιο, ο Επιτροπός Χόγκαν, είπε ότι θα επανέλθει για το θέμα αυτό τον Ιούνιο και νομίζω ότι θα είναι έτοιμα και τα συμπεράσματα της Προεδρίας ε, την ίδια εποχή. Γιατί μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για πιθανά περιθώρια από τον προπολογισμό 2016, περιθώρια τα οποία ούτως ή θα είναι σημαντικά. Δεν απέκλεισε όμως ο επίτροπο ένα πιθανό οικονομικό κίνητρο, συμπληρωματικό αυτών των τα οποία θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να προσφέρουν με το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων. Επίσης υπάρχει το αποθεματικό κρίσεως. Σε περίπτωση κρίσεως πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την αξιοποίηση του αποθεματικού κρίσεως. Για το 2016 είναι αργά. Πιστεύω ότι είναι αργά αν δεν βελτιωθεί όμω η κατάσταση την επόμενη χρονιά, πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και συμφωνώ κύριε Γιώργο σα, ότι τα λεφτά αυτά από τον ίδιο το Γεωργό προέρχονται. Όμω υπάρχει ο μηχανισμό, υφίσταται ο μηχανισμός και αν σε κάποιου τομεί βλέπουμε πιέσει μεγαλύτερε από ό,τι σε κάποιου άλλου, ίσω σε κάποιου να μην υπάρχουν και καθόλου πιέσει, η συζήτηση πρέπει να γίνει για την αξιοποίηση του, των πόρων αυτών. Και βεβαίω αυτά είναι συνέπειε αποφάσεων που ελήφθησαν ύστερα από μακρές συζητήσεις για μία πρόοδο προς μία κοινή γεωργική πολιτική προσανατολισμένη προς τις δυνάμεις της αγοράς με λιγότερη δύναμη ως προς τις ρυθμιστικές μας εξουσίες σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που ίσχυε στο παρελθόν. Βέβαια δεν είναι όλη αυτή η εικόνα και ο Επίτροπος Χόγκαν έχει αναλάβει δραστηριότητε και σε άλλους τομείς. Ξέρετε υπάρχει αυτή η αγορά, αυτή η task force, η ομάδα κρούσεως για τα για την αγορά γεωργικών προϊόντων και κυρίως εξετάζει τα διαρθρωτικά προβλήματα στο γαλακτοκομικό φορέ. Τομέα. Νομίζω ότι ο κύριος Γιάρη είπε ότι υπάρχουν αυτά τα ε, ε δυσνόητα, αυτές οι δυσνόητες συνθήκες, αυτή η ασυμβατότητα ε, μεταξύ του ενός και του άλλου δραστηριοποιούμενου στο γαλακτοκομικό τομέα. Όντως και με κάθε σεβασμό για τον γαλακ το κομικό τομέα και τους γαλακτοπαραγωγούς σε ορισμένε χώρες είναι μάλλον παραδοσιακή εμπνεύσεως. Οι γαλακτοπαραγωγοί δεν αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικές για μια καλή και σύγχρονη επιχείρηση εν έτη 2016 και συμφωνώ ότι δεν μπορεί ο Ευρωπαίος ε, ρυθμιστής και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνη της να δώσει λύσεις στα πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε, Άμεσες ενισχύσεις υπάρχουν και για το γαλακτοπαραγωγό που έχει γη στην ιδιοκτησία το έχουμε κοιτάξει τα στοιχεία και αυτή είναι σημαντική μίζων συμβολή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την επιβίωση των ε, γαλακτοπαραγωγών. Τα γνωρίζετε βέβαια όλα αυτά. Εγώ ήθελα απλώς να σας δώσω μια πιο, πιο ε, ε, ευρυγόνια εικόνα της κατάστασης. Κύριε Μαγκίνες, βελτίωση μέχρι αυτό το φθινόπωρο δεν βλέπω για την κατάσταση. Άρα πρέπει να οπλιστούμε για τις αγορές που αναφέρατε για ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο. Και νομίζω μπορώ να περάσω στα Ολλανδικά, κυρία Σράιερ. Με ρωτήσατε εάν ε, μπορούμε να ε, ρυθμίσουμε τα προβλήματα τα σχετικά με τα αζωτούχα και τα θείουχα κατάλοιπα. Ναι, υπάρχουν ανώτατα επίπεδα, το έχουμε παληθεύσει και με τις ελληνικές αρχές. Πρέπει να υπάρχουν ανώτατα επίπεδα και να τηρούνται αυτά στο γάλα. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου αρνητική. Η παραγωγή γάλακτος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την κατάργηση των ποσοστώσεων και νομίζω ότι και εδώ μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει ε, φτάσει το μήνυμα από τις αγορές στον τομέα. Να το επίπεδα τώρα για τις ε, τιμές σε θείουχα και αζωτούχα οφείλονται στο γεγονός ότι οι κατοχωρές για μακρό διάστημα δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές που αφορούν τα σχετικά, τη σχετική περιεκτικότητα του γάλακτος. Για το ρωσικό εμπάργο κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρση του εμπάργου και μέσω του οργανισμού, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που ξέρετε ότι μια απόφαση αναμένεται με πολύ θετικά συμπεράσματα ως προς τις την ευρωπαϊκή επιχειρηματολογία, αλλά και με, την, με τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουμε αναπτύξει. Βέβαια αυτά όλα γράφονται σε ένα πολύ ευρύτερο ε, πλαίσιο των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Ήταν τα επίπεδα επέμβασης και το βούτυρο με τις ερωτήσεις του κ. Ντες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το βούτυρο. Το επίπεδο είναι 5.000 στον αυτή τη στιγμή και δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση ακόμη. Άρα το πρόβλημα είναι η αποκορυφωμένη σκόνη γάλακτος και εκεί διπλασιάστηκε το, το επίπεδο, το, το όριο. Και έτσι έχουμε το περιθώριο μέχρι τις 180.000 τόνους να αγοράζουμε σταθερές τιμές. Για τα οπαρολαχανικά, Η Επιτροπή, κυρία Αγγιλέρα και κύριε Σεβαστιά, δεν θέλει κενό ανάμεσα στον ισχύοντα κανονισμό και τον νέο θέλει να το αποφύγει αυτό, άρα επεξεργαζόμαστε ένα νέο κανονισμό που θα πρέπει να τεθεί ενισχύ την 1η Ιουλίου και ενώ ο χάσμα δηλαδή πρέπει να υπάρξει. Αλλά σε αυτό θα χρειαστεί και η βοήθεια τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. Ε, αναζητούμε νέα προϊόντα γιατί υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν. Υπάρχει μια κάποια δυσφορία από ό,τι βλέπω από τους βουλευτές ότι ε, κινείται με, το, με ρυθμούς βραδύς η Επιτροπή, ότι δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να δεχθώ τέτοιες επικρίσεις, ε, τις άκουσα, σας βέβαια ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα μπορούσα βέβαια να σας δώσω κατάλογο όλων των μέτρων που έχουν εισαχθεί από το Αύγουστο του 2014 με την εισαγωγή του ρωσικού εμπάργου, τα πρόσθετα κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, δυστυχώ με τα 420 εκατομμύρια ευρώ που αποδεσμεύτηκαν το προηγούμενο Σεπτέμβριο για την προσαρμογή στην κρίση. Μόνο 192 εκατομμύρια δυστυχώ έχουν απορροφηθεί και δαπανηθεί από τα κράτη-μέλη, μόνο 45% του προπολογισμού που ήταν διαθέσιμος και νομίζω, Πρόεδρε, πως με αυτά τα τελευταία λόγια έδωσα απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόρτε. Δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε τη συζήτηση όλοι οι συνάδελφοι που ήθελαν να μιλήσουν μίλησαν, ακούσαμε τις απαντήσεις και μάλιστα όλος περίεργος ε, ολοκληρώνουμε και νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα. Αύριο συνεχίζουμε στις 9 το πρωί και θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες. Οπότε μην ξεχάσετε τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες ψηφοφορίες. Και ελπίζω ότι ο κύριος Σικέρσκι θα έρθει για να προεδρεύσει αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Χαίρετε.